Colleagues, good morning. καλημέρα. Να επαναλάβουμε την ε, συνεδρίαση. Πριν ε, ξεκινήσουμε, ο κύριος Μπράντμπερν ζήτησε τον λόγο τη της διαδικασίας. Φίλιπ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να θίξω ένα γενικό ζήτημα, δεν αφορά μόνο την Επιτροπή μας αλλά προέκυψε χτες στην Επιτροπή μας, οι βοηθοί μας μετακινούνται για να καθίσουν ε, άνθρωποι από άλλα θεσμικά όργανα. Ε, όσον με αφορά, και αυτό δεν αφορά μόνο το δικό μου βοηθό, είναι ζωτικό το έργο τους ε, για τη δουλειά μας, παρακολουθούν τις εργασίες μας, σημειώνουν και μας βοηθάνε πάρα πολύ είναι οι δεύτεροι πιο σημαντικοί άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα. Ε, οι υπόλοιποι πλην της γραμματείας είναι διακοσμητικοί εδώ μέσα. Οπότε αν υπάρχει έλλειψη χώρου θα επιμείνω κανένας βοηθός να μην σηκώνεται από τη θέση του κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης. Thank you, uh, I, I know had a particular problem this week. Your, well made. because Έχετε δίκιο και όπως θυμάστε έχουμε ήδη αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και στο παρελθόν. Η αίθουσα αυτή είναι μικρή, δημιουργούνται προβλήματα. Σημειώνω αυτό που είπατε επειδή δεν ήξερα ακριβώς ποιο ήταν το θέμα σκέφτηκα ότι θα μπορούσατε να έχετε το δικαίωμα απάντησης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τους ε, κλητήρες να είναι πιο ευαίσθητοι στο θέμα των βοηθών ειδικά όταν είμαστε σε αίθουσες όπου δεν υπάρχει πολύ χώρος. Αν έχουμε μεγάλη αίθουσα στη διάθεσή μας δεν υπάρχει πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα. We now go on uh, Περνάμε στις ψηφοφορίες, αν είστε έτοιμοι. Έχετε τις κάρτες σας. We'll, I'm going to do a test first. Do you think you could get your... Μια δοκιμή πρώτα. Κύριε Ντεβερά, η κάρτα σας στο Στρασβούργο. Θα σας πάρει λίγη ώρα να πάτε να την βρείτε από το Στρασβούργο. Has everybody got their cards apart from Mrs. De Verac? Εκτός από την κυρία Ντεβεράκ, οι υπόλοιποι έχετε τις κάρτες σας. Ωραία, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Κύριος Αλκαντράουι, έρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν 25, 21 υπέρ, 4 αποχές, κανένας κατά. Άρα εγκρίνεται το ότι έχετε υπέροχο πρόεδρο. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε. Έκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την αλλαγή του κλίματος. Παράγραφος 1, τροπολογία 3, Άουκεν. Υπέρ. Συγγνώμη, κυρία Άουκεν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 6. ένα λόβα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε, ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν 28. Ναι, η κυρία Ντεβεράκη είναι κατά. 15 υπέρ, 13 κατά, μία αποχή εγκρίνατα. Οι 7 καταπίπτει, όχι, συγγνώμη, μόνο το δεύτερο μισό. Ψηφίζουμε το πρώτο μισό της τροπολογίας 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 Μαρινέσκου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία Α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει. Στις 9 ψηφίζουμε πρώτα το πρώτο τμήμα. Μέχρι τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο υπέρ, κατά, αποχές, εγ... απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Συμβιβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα Καταπίπτει 36. 12 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Στην 4α παράγραφο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Κυρία Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 για την παράγραφο 4β υπέρ, κατά, άποχες. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Τροπολογία 16. Τι κάω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 17 κατά και μία αποχή απορρίπτεται λοιπόν. Η 17 αποσύρθηκε, η 18 βλάστο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 για την 5α νέα υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 20 και 21 καταπίπτουν. 22 κυρία Τικάου. Έχουμε μια προφορική τροπολογία εδώ. Κυρία Τικάου παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά την κοινή θαλάσσια πολιτική βάζουμε το που λαμβάνει υπόψη which takes into due account που λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν διαφωνίες επί της προφορικής τροπολογίας. Αν όχι, τότε ψηφίζουμε την 22 με την τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 5β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την παράγραφο α 25 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Παράγραφος 6β, τροπολογία 27 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Συμβιβαστική γάμα για την παράγραφο 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29-32 καταπίπτουν. Πάμε στην παράγραφο 7α νέα. Τροπολογία 33. Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 και 36 καταπίπτουν η 37 για την 7β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την παράγραφο 8α, προφορική τροπολογία για την τροπολογία Βλάστο. Θα τη διαβάσετε παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να προσθέσουμε στο τέλος μετά το υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η εκστρατεία πληροφόρησης και λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των κρατών μελών κτλ. Έγινε κατανοητή η προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 1. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι το is increasing υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μόνο το πρώτο τμήμα έγινε δεκτό τροπολογία 2 για την ιδεολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 33, 34 με την κυρία Ντεβεράκ. 32 υπέρ, 2 αποχές. Καμία ψήφος κατά. Α, έχετε την κάρτα σας τώρα. Άρα 31 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. The next item on Το επόμενο σημείο είναι οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία. Η ο κύριος Στέρεξ. Περιμένουμε λίγο να φύγουν ορισμένα άτομα και Θα δώσω τα ενία στον Αντιπρόεδρο για να πάω στην Επιτροπή Γεωργίας. Ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος δεν θα μας αφήσει για πολύ χρόνο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Στέρξ για την παρουσίαση της έκθεσής τους σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά το κατάπλου και απόπλου απολυμμένα στο κρατών μελών της κοινότητας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ πέρα πρόκειται κατ' ουσίαν για μια ανακοίνωση της Κομισιόν, ένα σχέδιο δράσης και μια πρόταση οδηγίας. Στην ανακοίνωση η Κομισιόν εξηγεί πώς θέλει να ενθαρρύνει την ε, ναυτιλία με το να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια εντός της ε, κοινότητας όσον αφορά τις μεταφορές κάνει διάκριση μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέτρων και υπάρχει ένα πρώτο βήμα που πρέπει να δημιουργηθεί μέχρι τις 2010 ε, με απλοποίηση κανόνων και λογικά, μετά μέσω μακροπρόθεσμα μέχρι το 2013 και μετά γίνονται κάποιες συστάσεις ε, στα κράτη-μέλη που πρέπει να ολοκληρωθούν ε, μέχρι το 2020. Υπάρχουν ε, κάποιοι πρακτικοί λόγοι για την ε, εφαρμογή αυτής της οδηγίας γιατί έχουν προκύψει άλλα έγγραφα από τον IMO οπότε έχει αλλάξει κατάσταση και όσον αφορά τους κανόνες ασφαλείας. Έχουμε επίσης επιβεβαιώσει πως πλέον ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο η ψηφιοποίηση των πληροφοριών και ανταλλαγή, και τους μεταξύ λιμένων και κρατών μελών οπότε με την πρόταση αυτή η Κομισιόν λέει πως πρέπει να συμπληρώνουν όλα τα διεθνή έγγραφα, όλα τα κράτη-μέλη. Μετά το net, το οποίο αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και την επιτήρηση την αυσιπλοείας, πρέπει να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο ε, στο οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίε για τα φορτία Μέσω αυτού του συστήματος δηλαδή πρέπει να συμβαίνουν τα πάντα και για αγαθά τα οποία παραμένουν εντός της ε, κοινότητας δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνονται και να παραδίδονται τα έγγραφα γιατί είναι κάτι το πολύ απλό πλέον όπως με τα φορτηγά και δεν, χρειάζεται, δεν χρειάζονται όλες αυτές οι διατυπώσεις. Νομίζω πως πρόταση Κομισιόν είναι καλή πρόταση και πράγματι πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, ναυτιλία γιατί υπάρχουν ε, ε, περιοχές που μπορούν να ωφεληθούν πάρα πολύ όσον αφορά τις μεγάλης απόστασης μεταφορές καθώς πρόκειται και για μια μεταφορά φιλική προς το περιβάλλον και σε σύγκριση με τα φορτηγά έχει κάποιες εντυπώσει παραπάνω οι οποίε δεν χρειάζονται. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω τώρα κάποια πράγματα στην πρόταση της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα ε, δεν μιλάμε μόνο για απλοποίηση αλλά και για εναρμόνιση. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερον, και αυτό θα το βάλω και στην έκθεση, το θέμα δεν είναι μόνο διοικητικές υποθέσεις σε σχέση με τις ε, μεταφορές. Αφορά και τα τελωνία, κάτι το οποίο είναι ίσως πολύ σημαντικότερο ε, σε αυτό το κομμάτι από τι μεταφορές. Επίσης υγειονομική έλεγχη, φύτεο υγειονομική έλεγχη και όλα αυτά και ασφάλεια. Στην περίπτωση στην οποία ε, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα ε, μαζί και ταυτόχρονα νομίζω θα έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Αλλά εάν δεν απλοποιηθούν τα τελωνία τότε το πρακτικό αποτέλεσμα ε, είναι λιγότερο αισθητό για εμάς στην πράξη. Οπότε θέλω να αναφέρω και στην έκθεση πως Δεν μπορούμε βέβαια να επηρεάσουμε τα πράγματα όπω θα θέλαμε θεωρητικά, αλλά εδώ πέρα απευθύνομαι κυρίω στην Κομισιόν και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό στην Κομισιόν και το Συμβούλιο, πω ε, τα διαφορετικά τμήματα του μηχανισμού της Κομισιόν ε, και των κρατών μελών πρέπει να καταλήξουν σε μια λύση η οποία θα είναι πραγματική λύση. Ένα τρίτο νομίζω σημείο, εν πάση περιπτώσει το επόμενο σημείο, είναι ένα δύσκολο σημείο στο Συμβούλιο, όχι τόσο στο Κοινοβούλιο, η χρήση μίας κοινή γλώσσας. Η πρότασή μου είναι σαφή σε μένα. Νομίζω πως τα αγγλικά πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως γίνεται και στην αεροπορία. Και όπως γίνεται ήδη στην αυτιλία σε μεγάλο βαθμό. και νομίζω πρέπει να μπορέσουμε να γράψουμε κάτι τέτοιο και στους δικούς μας ε, κανόνες. Ε, το SAFES είναι ένα σύστημα επίσης το οποίο υπάρχει, έχει πάρει βραβείο από την ΕΜΣΑ στην ε, Λισαβόνα. Περιέχει όλες τις πληροφορίες. Επίσης έχω προσθέσει μία πρόταση για την πρόσβαση στα στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν έναν έλεγχο πρόσβαση, είναι ευαίσθητε εμπορικά πληροφορίε. Πρέπει λοιπόν να το ρυθμίσουμε αυτό, να αποφασίσουμε οι αρχέ, εν πάση περιπτώσει, ποιο έχει πρόσβαση και ποιο δεν έχει και να φροντίσουμε να υπάρχει πραγματικά επιτήρηση αυτού του πράγματο. Τώρα για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων. Υπάρχουν ε, κάποιοι άνθρωποι από την πραγματική ζωή, θα το έλεγα έτσι, που το ερμηνεύουν αυτό με διάφορους ε, τρόπους. Δηλαδή λένε πως το fax δεν είναι ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Οπότε ξεκαθάρισα κάπως τον ορισμό για να ξέρουμε με ποιο σύστημα και με ποιο τρόπο πρέπει να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες. Επίσης, ε, ναι το είπα αυτό, απαλλαγή των πληροφοριών, ε, απλοποίηση των εντύπων. Ε, τώρα για τα μέσο πρόθυμα ή τα μακροπρόθυμα, δεν θυμάμαι μέτρα, στις συστάσεις εκεί πέρα όπου μιλάμε για την υπηρεσία πλοήγησης ε, όπου θα πρέπει να υπάρξει μια πιο έγκαιρη ειδοποίηση και να μπορέσουμε να την οργανώσουμε καλύτερα για να μπορούν ε, τα πλοία να, να μπαίνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια γιατί το βάρος δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά συχνά είναι και διαδικαστικό και θα μπορεί π.χ. να πάρει το δίπλωμα πλοηγού ο καπετάνιος ε, καθώς ε, συχνά είναι πάρα πολύ υψηλέ οι προδιαγραφές για να συμβεί κάτι τέτοιο. Γνωρίζω πως ε, δεν θέλουν να τα ακούσουν κάτι τέτοιο τα, τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω εγώ πως είναι σημαντικό. Στην περίπτωση δηλαδή στην οποία ο καπετάνιος με το πλοίο του μπαίνει συνέχεια σε ένα λιμάνι, το γνωρίζει ε, και μπορεί δηλαδή να τον εξετάσουμε και να δούμε εάν έχει την ικανότητα να πλοηγήσει το πλοίο του και να μην χρειάζεται να περιμένει τον πιλότο να ανέβει πάνω. Επίσης θα ήθελα να μην δούμε μόνο τη σύνδεση ανάμεσα στη θάλασσα και το λιμάνι αλλά και το τι γίνεται παραμέσα στην ενδοχώρα την ε, σύνδεση δηλαδή και ειδικά όσον αφορά βεβαίω ε, την εσωτερική ναυσιπλοεία για τη μετάβαση από την ε, ποντοπόρο ναυτιλία στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Το τι μπορεί να γίνει για να γίνει και γρήγορα κιόλα κάτι τέτοιο, να υπάρξει μια σύνθεση, να φέρει γρήγορα η Κομισιόν κάποιες προτάσει για να υπάρξει π.χ αυτό το δίκτυο πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλογίας, το οποίο πρέπει να συνδεθεί με το net για να επιταχυνθούν ορισμένα πράγματα γιατί πράγματι πολλά λιμάνια δεν ε, σκέφτονται καθόλου τη σύνδεση με την ενδοχώρα και τέλος η προθεσμία στην πρόταση της Κομισιόν 2013 πρέπει να τη διατηρήσουμε νομίζω γιατί είναι και μεγάλες οι, οι επενδύσεις. Νομίζω πως είναι ρεαλιστική και η Κομισιόν Και δεν είμαι τώρα υπέρ της τακτικής να προτείνουμε μία άλλη ημερομηνία για να διαπραγματευτούμε, να γίνει 2013, αλλά όντως να ισχύσει 2013. Αντιλαμβάνομαι πως αυτή τη στιγμή ε, φεύγουμε από την οικονομική κρίση και περνάμε σε μια ανάπτυξη οπότε θα ξαναρχίσει βεβαίως ε, η άξη της οικονομίας και των μεταφορών και θα οδηγηθούμε ξανά στα ίδια τα προβλήματα οπότε πρέπει να σταθεί στα πόδια του και να λειτουργεί αυτό το σύστημα να επενδύσουν τα λιμάνια Και βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο θα ζητάνε οι παράγοντε συναθλίε, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν οι αρχέ. Και ελπίζω βεβαίω να με στηρίξουν οι συνάδελφοι στην κατεύθυνση αυτή και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ κύριε Στέξ. Πραγματικά εξαίρετη η ποιότητα της έκθεσής σας. Και είχατε και το θάρρος να παρουσιάσετε τις απόψεις σας και να δείξετε και έναν μεταδοτικό, μια μεταδοτική αισιοδοξία για την κρίση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντανές Πασκουάλ. Πώς λέγεται. Στο σκιώδη Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητή συζήτησε τη στήριξή μας και δίχως άλλο θα την έχει. Η έκθεση αυτή, κατά την άποψή μας, είχε πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Αυτή ήταν η αρχική μας εντύπωση, την οποία τώρα επιβεβαιώνουμε. Εργάστηκε ο εισηγητής με το συνήθι τρόπο εργασίας, μίλησε με όλους τους ενδιαφερόμενους, μίλησε με τους σκιώδεις εισηγητές, βεβαίως με μένα και δημιούργησε ένα σύστημα ακροάσεων όπου οι πραγματικοί ειδικοί, αυτοί που βιώνουν καθημερινά το θέμα, κατάφεραν να μας εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους. Πρόκειται για μια πληρέστατη έκθεση Είχα ορισμένε ανησυχίε, τις οποίες τις εξέφρασα στο παρελθόν. Οι ανησυχίε αυτέ, οι προβληματισμοί ελήφθησαν υπόψη σε αρκετέ από τι τροπολογίε ιδιαίτερα σε αυτή που φοράει το άρθρο 7α σχετικά με τι ευαίσθητε πληροφορίε. Πιστεύω ειλικρινά ότι πρόκειται για κανόνε που θα μπορούσαν να εξυγχρονίσουν το σύστημα επικοινωνιών, αποφεύγουν τη γραφειοκρατία, είναι πραγματικά θαραλές και ελπίζουμε ότι εξίσου ρελέω με το Κοινοβούλιο να αποδειχθεί και το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να αναμένετε μερικές δυσκολίες από πλευράς του Συμβουλίου, γιατί δίχως άλλο θα υπάρξουν αντιστάσεις στην ιδέα ε, του, το, της χρήσης των αγγλικών γιατί είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται από την αυσιπλοεία. Θα πρέπει όμως να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε τα αγγλικά να είναι η κοινή γλώσσα αλλά να προβλέπονται και ορισμένες εξαιρέσεις για ορισμένες δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να επαναλάβω ότι σαφώς είμαστε υπέρ αυτής της έκθεσης. Λέτε ότι είναι τεχνική αυτή η έκθεση Βεβαίως και είναι. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πρόβλημα διαλεκτικής και αντιπαράθεσης διαφορετικών απόψεων που στην ουσία εδώ δεν υπάρχουν. Εδώ κατά βάση πρόκειται για την λήψη μιας σοβαρής και θαραλέας πολιτικής απόφασης. Αν καταφέρουμε να την πάρουμε θα εξυγχρονιστούν πολλά συστήματα. Συνεχίστε Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μα. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω θα τα σκόπιμο να υποβάλουμε τροπολογίε, δεν νομίζω. Αν είναι αναγκαίο όμω θα το κάνουμε. Ενδεχομένω θα διοτυπωθούν ορισμένε αφιβολίε από ορισμένα άλλα μέλη του Κοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, εμεί θα συνεργαστούμε μαζί σα έτσι ώστε να τύχει κάθε στήριξη αυτή, η έκθεση. Ο κ. Δηλάνα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, κ. Πασκάλ. Εμείς σήμερα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ καλή κοινοποίηση και έγκαιρη κοινοποίηση της Επιτροπής και μια πολύ καλή δουλειά του εισηγητή. Θα έπρεπε λοιπόν να μην το συζητήσουμε καν το θέμα. Τι εννοώ ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής γίνεται πολύ έγκαιρα σε σχέση με τα όσα παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με αυτό το τομέα. Και αυτό το κάνει εντάσσοντα την ανακοίνωση αυτή στα πλαίσια μια άλλη ανακοίνωση που αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο Θαλασσίων Μεταφορών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αποτελεί σημαντική ψηφίδα αυτής της ανακοίνωση. Το είπε και ο άλλο κοιόδη εισηγητή. Ο εισηγητή είπε ήταν ε, πραγματικά άψογος και σε ό,τι αφορά ε, τη σχέση μεταξύ των βουλευτών, μεταξύ των ομάδων. Πήραμε μέρος ε, στις ακροάσεις. Εξετάστηκαν με πολύ προσοχή όλες οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν και παράλληλα θα μας κεράσει ένα καφέ μετά, εντάξει. υπήρξε αντικειμενικά και η ικανότητα να παρουσιαστούν περιληπτικά οι διάφορες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. Πιστεύω ότι με θετικό τρόπο ερμηνεύτηκε αυτή η υπόδειξη που έγινε σχετικά με την ενσωμάτωση αυτής της ανακοίνωσης ως σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των θαλασσίων μεταφορών ή να προωθηθεί και η ιδέα των ε, μεταφορών σε, ποτάμι, σε ποτάμια. γιατί αυτή η πρόταση οδηγίας είναι πολύ σημαντική. Περνάει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα πρέπει να οθήσουμε την Επιτροπή να ασχοληθεί και με άλλα θέματα, όχι μόνο με τις χερσαίες μεταφορές. Σήμερα περιοριζόμαστε στο να αναφέρουμε ένα σχέδιο απλοποίησης, εναρμόνισης. Προτείνουμε οι μεταφορές αυτές να ενταχθούν εδώ, αλλά πιστεύω ότι για τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πλαίσιο και να καλέσουμε την Επιτροπή να συμπληρώσει αυτή την επιχείρηση. Πάρα πολύ συχνά ε, δεν εκτελονίζονται τα εμπορεύματα στους λιμένες ε, ε, εκτελονίζονται στην ενδοχώρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε έτσι ώστε η Επιτροπή θα καταφέρει να εξετάσει και άλλες φάσεις της πορείας που ακολουθούν τα εμπορεύματα. Μία μικρή παρατήρηση σχετικά με το άρθρο 3. Το άρθρο 3 αφορά τον ορισμό των συστημάτων που αφορούν την ηλεκτρονική μεταβίβαση των δεδομένων. Δεν γνωρίζω αυτά τα λειτουργικά, τα προγράμματα. Είναι προγράμματα διαχείρισης των συστημάτων. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια υπόδειξη, όχι μια ξερή δήλωση. Για την ώρα δεν γνωρίζω αν στις διάφορες χώρες υφίσταται η απτή δυνατότητα στα σημεία κατάπλου να ενταχθούν αυτά τα σημεία. Και πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια δισκαμψία. Δεν θα ήθελα αύριο κάποιος να υποβάλει ένα άλλο πρόγραμμα, ο Bill Gates τη στιγμή που θα μας δώσει κάτι ακόμα πιο συγκεκριμένο, ακόμα πιο απλοποιημένο που θα γίνει η κοινή γλώσσα, όπως στην ουσία είναι τα γλυκά τώρα. Αυτό θεωρήστε το μια περιθωριακή παρατήρηση επί της οποίας ήταν σκόπιμο να σκεφτούμε. Πιστεύω ότι ο συγητή έχει εμπαθύνει πολύ περισσότερο από εμά, αλλά επιτρέψτε μου απλά και μόνο να διατυπώσω αυτή τη σκέψη. Και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ε, ότι έχω στοιχεία για να πω ότι θα πρέπει να, γίνουν, να υποβληθούν περαιτέρω τροπολογίες. Ο εισηγητή με πάρα πολύ ακριβή τρόπο έλαβε υπόψη του όλες τις παρατηρήσεις, κατάφερε να τις ε, εντάξει και να τονίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα γιατί μολονότι κρίνεται πολύ καλή η εργασία της Επιτροπής οι υποδείξεις που υποβάλλουμε είναι υποδείξεις χρήσιμες για την Επιτροπή και ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα της σχέσης που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ ημών και της Επιτροπής. Εγώ είμαι πολύ λιγότερο απεσιόδοξο σε ό,τι αφορά τις απόψεις του Συμβουλίου διαπιστώνω ότι υπάρχει ανάγκη παρέμβασης και από πλευράς Συμβουλίου. Δεν θα έλεγα ότι είμαι απεσιόδοξο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν μάχες σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο. Το θέμα είναι λιγάκι η χρόνη εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αυτό θέμα, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει αυστηρά να τηρήσουμε τη γραμμή που επιλέξαμε. Και αυτό σε ό,τι αφορά μερικά από τα στοιχεία που θα μπορούσαν άμεσα να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων θα ήθελα να πω στον κύριο Στέξ ότι συμφωνούμε με τα ουσιώδη σημεία της έκθεσής του και σε ό,τι αφορά το πνεύμα και σε ό,τι αφορά το γράμμα. Πραγματικά, λαμβάνει υπόψη το στόχο της Επιτροπής που αφορά την ορθολογικοποίηση και απλοποίηση της ναυσιπλοείας και αυτό το επιτυγχάνει χάρη στις παρατηρήσεις και χάρη στις τροπολογίες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των διαδικασιών που κατά την άποψή μας είναι ένας ε, στόχος ιδιαίτερα σημαντικός πέρα από τις τεχνικές πτυχές του. Θα ήθελα ιδιαίτερα να χαιρετήσω τις προσπάθειες που κατέβαλε ο κύριος Στέρξε σε ό,τι αφορά τον ιστορικό ορίζοντα, δηλαδή το 2013 το 2013 ε, ε, δεν θα πρέπει να είναι κάτι αφηρημένο. Θα πρέπει να εκφράσουμε την πραγματική βούληση να εφαρμόσουμε τα όσα περιέχονται εδώ. Εμείς ε, θα θέλαμε να τον συγχαρούμε, όχι για τεχνικούς λόγους, γιατί πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Πιστεύουμε ότι η προώθηση αυτού του τρόπου θαλασσίων μεταφορών είναι λιγότερο, ε, περισσότερο ασφαλής, περισσότερο οικολογική και νομίζω ότι κινούμεθα προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί λαμβάνονται οι υπόψη οι οικολογικοί προβληματισμοί που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε. Θα έκανα παρόλα αυτά δύο παρατηρήσεις για την έκθεση του κυρίου Στέρξε. Αυτό αφορά τη γλώσσα που μιλάμε και τη γλώσσα την πληροφορική. Εμείς ε, που είμαστε σαφώς υπέρ της πολιτιστικής διαφοράς των λαών και της διαφοράς των γλωσσών Υποστηρίζουμε παρόλα αυτά την αρχή που υποστηρίζεται, την αρχή δηλαδή με κοινή γλώσσα για την επικοινωνία στον τομέα της επικοινωνίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτή την εναρμόνιση, θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή γλώσσα και κατά την άποψή μας η χρήση των αγγλικών δεν ε, συνεπάγεται την εγκαθίδρυση μιας δικτατορίας μιας γλώσσας και δεν ε, οδηγεί στην διακύβευση των άλλων γλωσσών. Παρόλα αυτά, για να λάβουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και μία άλλη πραγματικότητα. Τα αγγλικά δεν είναι μία συνήθις γλώσσα στους μικρούς ε, λιμένες. Θα προτείναμε να επεκταθεί το μέτρο για την κοινή γλώσσα για τους μικρούς λιμένες έτσι ώστε να φτάσουμε σε συγκεκριμένα μέσα σε συγκεκριμένες διαδικασίες που θα επιτρέπουν μία πιο ήπια εισαγωγή αυτού του μέτρου. Δεύτερη παρατήρηση σχετικά με την γλώσσα της πληροφορικής και το ηλεκτρονικό σύστημα μεταβίβασης δεδομένων. Μας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα θετική ιδέα η κοινή γλώσσα, ε, ότι η κοινή γλώσσα θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια μεγαλύτερη ε, εναρμόνιση. Θα πρέπει όμως να ασχοληθείτε περισσότερο με θέματα συμβατότητας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των ήδη υπαρκών των συστημάτων μεταβίβασης δεδομένων. Οι δύο αυτές έχουν στόχο την εισαγωγή μιας μεγαλύτερης ευελιξία στις νέες αυτές διαδικασίες έτσι ώστε να μην ε, δημιουργηθεί μια βάση για το διαδεδομένο συνέστημα μεταξύ των Ευρωπαίων ότι δηλαδή μας επιβάλλονται νέοι περιορισμοί και με τρόπο πάρα πολύ απότομο. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους ε, της ομάδας μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στίρξ, τον εισηγητή, ο οποίος ε, έκανε πολύ καλή οργάνωση του θέματος. Είχαμε και ένα μίνι σεμινάριο που επέτρεψε στους σκιώδεις εισηγητές να συζητήσουν με εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία, κάτι που θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο για όλους μας. Τώρα για την έκθεση. Αρχικά ήμασταν πεπισμένοι ότι το έργο μας δεν θα ερχόταν σε σύγκρουση με διεθνείς συμφωνίες και προχωρήσαμε με αυτή τη λογική. Οι τροπολογίες είναι πολύ καλές. Θεωρώ ότι η τροπολογία 23 είναι ιδιαίτερο καλή γιατί θέτει το θέμα της εσωτερικής αγοράς και τη στηρίζουμε. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων και την ε, ημερομηνία έναρξής της. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη συγκεκριμένη προθεσμία, όμως έχουμε κάποια προβλήματα με τις ε, σύντομες μεταφορές. Γενικά όμως θεωρούμε ότι η ημερομηνία είναι λογική, απλά θα πρέπει να δούμε αν όλοι μπορούν να συμμορφωθούν με αυτή. Ένα άλλο θέμα που θέσαμε στους εμπειρογνώμονες και δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Στέρξ μπορεί να με βοηθήσει εδώ. Μιλούσαμε για τα κράτη-μέλη και αναφέρθηκαν ότι μπορεί να έχουμε φορτίο σε ένα εμπορευματοκιβώτιο που προέρχεται και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν μέρει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται με αυτό το εμπορευματοκιβώτιο. Αν και από ό,τι κατάλαβα θα είναι εύκολο να γίνει η διάκριση με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα και χαίρομαι που άκουσα τον συνάδελφο να μιλάει για κοινή γλώσσα. Είναι ωραίο να ακούμε κάποιον που έχει μητρική γλώσσα τα αγγλικά. Όμως δεν πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί εδώ. Στην βιομηχανία της αεροπορίας διεθνώς χρησιμοποιούνται τα αγγλικά. Όμως όταν μιλάμε για μικρά μέρη ή για τον τοπικό εναέριο χώρο υπάρχει ευελιξία. Το θέμα αυτό είχε προκύψει και στο σεμινάριο του κυρίου Στέρεξ. Αλλά, για παράδειγμα, εγώ είχα πάει διακοπές κρουαζιέρα και γενικά ομιλή μιλούσαν αγγλικά, αλλά τους ρωτούσα τι κάνετε όταν βρίσκεστε σε ένα μικρό λιμάνι και πρέπει να συνεννοηθείτε με τους αλληλείς οι οποίοι ενδεχομένως δεν μιλάνε αγγλικά και γενικά από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ευελιξία και συνήθως φροντίζουν να έχουν κάποιον ο οποίος μπορεί να συνεννοηθεί στην τοπική γλώσσα. Είναι δηλαδή ρεαλιστές σε αυτό το θέμα γιατί το σημαντικό είναι η ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει και ο κύριος Στέρξ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έθεσαν ενδιαφέροντα θέματα. Θα στηρίξουμε την έκθεση και ελπίζω ότι θα προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Κύριε Στέρξ, από ό,τι φαίνεται πάει καλά σε μία όχι τόσο εύκολη έκθεση. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στέρξ για την ενδιαφέρουσα έκθεσή του. Ε, λέγοντας βεβαίως πως μου αρέσει και εμένα ο καλός καφές όπως ε, ζήτησε και ο συνάδελφος, αλλά έχω κάποια πράγματα να ρωτήσω. Όταν μιλάμε για τα δεδομένα των φορτίων, έχουμε το σύστημα αυτόματης ε, αναγνώρισης των φορτίων, το AIS, όπου υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που αφορούν το φορτίο για λόγους ασφαλείας. Πιθανόν λοιπόν μπορούμε να μεταδώσουμε αυτά τα δεδομένα όσον αφορά το φορτίο και για την ε, εκφόρτωση του φορτίου. Να τα μεταδώσουμε λοιπόν. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι και προς την Κομισιόν τι ρόλο θα παίξει το Γαλιλαίο και στο μέλλον και αν ε, θέσουμε ως όριο το 2013 θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εντατικά το Γαλιλαίο ως σύστημα πλοήγησης και πληροφοριών στην Ευρώπη. Το δεύτερο ερώτημα Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να απλοποιηθεί πράγματι το σύστημα των πλοηγών. Γιατί πλοία τα οποία μπαίνουν συνέχεια στο ίδιο λιμάνι, καμιά φορά ο καπετάνιος ξέρει καλύτερα το λιμάνι από τον πλοηγό, αν ο πλοηγός είναι νέος στη δουλειά. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και να εξεταστεί βεβαίω ο καπετάνιος και να έχει μετά ένα γράμμα, ένα πιστοποιητικό κάτι, πώ δεν μου χρειάζεται οπωσδήποτε ο πλοηγός, ξέρω εδώ πέρα το λιμάνι, ξέρω την τάδε από βάθρα κτλ. Ε, πότε βλέπετε να, να το ξεκινάτε αυτό. Merci, ε, Ευχαριστώ. Κύριε Στέρξ, ε, σας ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι καταφέρατε να ισορροπήσετε μεταξύ φιλοδοξίας και ρεαλισμού. Κάποια πραγματάκια νομίζω με απασχολούν ακόμα. Ο κύριος Κούν μόλις τα ανέφερε, η πλοηγή συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, ότι δηλαδή πρέπει να προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες στον καπετάνιο, αν γνωρίζει καλά την περιοχή, να βάλει μόνο στο ίδιο στο πλοίο στο λιμάνι. Από την άλλη όμως θέλω να υπάρχει ο χώρος για ειδικά ύδατα τα οποία χρειάζονται πλοηγό και έχουν το χαρακτηριστικό ε, ότι υπάρχει άμμος η οποία μετακινείται από εδώ και από εκεί γρήγορα και από μέρα σε μέρα δυσκολεύονται και οι πλοηγοί να παρακολουθήσουν την αλλαγή στην ε, μορφολογία. Οπότε υπογραμμίστε το αυτό λίγο για αυτές συγκεκριμένες, ε, για αυτές συγκεκριμένες περιοχές. Ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πλοηγών. Τώρα για τη σύνδεση που γίνεται μεταξύ SafeSynet και River Information System, το δίκτυο πληροφοριών εσωτερική ναυσιπλοεία. πράγματι ενδιαφέρον αυτό, όπως και αυτό το οποίο λέτε πως πρέπει να υπάρχει μία γλώσσα και αυτή να είναι τα αγγλικά. Αλλά αν μιλάμε να γίνει σύνδεση μεταξύ του RIS και του SafeSynet, εγώ θα πήγαινα ένα βήμα ακόμη παραπέρα και θα έλεγα πως ε, και στην εσωτερική ναυσιπλοεία πρέπει να οδηγηθούμε σε μία γλώσσα. Και το λέω αυτό γιατί η σύνδεση μεταξύ ε, ναυτιλίας και εσωτερικής ναυσιπλοείας πρέπει να γίνει πιο έντονη και δεύτερη σκέψη είναι πως βλέπουμε πως και στην εσωτερική ναυτιλία έχουμε όλο και περισσότερους ναύτες που προέρχονται από χώρες με εξωτικές γλώσσες και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εισρωή Φιλιππινέζων στην εσωτερική ναυτιλία. Ε, το ξέρω ότι σας προκαλεί έκπληξη, αλλά είναι τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολύ μεγάλη εισρωή Φιλιππινέζων στα ποτάμια, ναι. Στην εσωτερική ναυτιλία. Οπότε ούτως ή άλλως έχουν επικρατήσει τα αγγλικά και ε, όπως ξέρετε κι εσείς υπάρχουν καμία φορά ατυχήματα που προκαλούνται από την ασυνεννοησία. Οπότε πρέπει ε, όταν θα γίνει η σύνδεση μεταξύ RIS και SafeSynet να περάσει και ε, μία γλώσσα στην ε, εσωτερική ναυτιλία. Θα μπορούσατε ίσως να το συμπληρώσετε. Αυτά από μένα κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα δύο συγκεκριμένα σημεία για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Eh Εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, θα δώσω το λόγο στον κύριο Στέρεξ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Η Επιτροπή μπορεί να πάρει το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστούμε και τους σκιώδεις εισηγητές και τους υπόλοιπους ε, ευρωβουλευτές για τα θετικά του σχόλια. Γιατί είχαμε αυτή την πρόταση. Ο εισηγητής έχει δίκιο αν ξεκινήσετε από τη Μαδρίτη για να πάτε τη Γερμανία δεν έχετε κανέναν έλεγχο. Αν κάνετε την ίδια διαδρομή μέσω μιας ε, άλλης χώρας ε, τότε έχουμε πολλούς ελέγχους και αυτό είναι προβληματικό αν προσπαθήσουμε να κάνουμε την ίδια διαδρομή μέσω πλοίου. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα για τα πλοία, κάτι που αφορά και τους τελωνιακούς κανόνες και τους κανόνες που έχουν να κάνουν με τους λιμένες κτλ. Πού βρισκόμαστε επί της διαδικασίας. Το Συμβούλιο έχει προσπαθήσει πολύ. Είχαμε πολλές ε, συνεδριάσεις με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας και κατέληξε στο τέλος του έτου σε μια κοινή θέση κατά κάποιο τρόπο την οποία διατηρήσαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να μην συμφωνούμε με όλα. Υπάρχει ένα θέμα ειδικά με το οποίο διαφωνούμε όσον αφορά τις καθυστερήσεις. Βεβαίως μας λένε ότι θα έπρεπε εν ώψη του 2020 και των αλλαγών λόγω κλίματος να υπάρξει καθυστέρηση. Δεν θεωρούμε ότι θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Καταρχάς, γιατί θα ξεκινήσει η λειτουργία του SafeSynet, κάτι που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και σας υπενθυμίζω ότι και ο οργανισμός μας, η ΕΜΣΑ, πρόκειται να βοηθήσει πολύ και επίσης θα έχουμε και τα ηλεκτρονικά τελωνία, τα e-customs από το 2013. Άρα θα έχουμε αυτές τις υποδομές. Βέβαια θα υπάρξουν κάποια προβλήματα με τα μικρά λιμάνια, αλλά συνήθως στα μικρότερα λιμάνια δεν έχουμε αυτού του είδους τις μεταφορές που μας ενδιαφέρουν στην πρότασή μας. Άρα θέλουμε να παραμείνει η ημερομηνία του 2013. Τώρα, ακούσαμε κάποια ενδιαφέροντα σχόλια από τους ομιλητές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην προσέγγιση του Συμβουλίου. Ίσως υπάρξουν δυσκολία για την αποδοχή ορισμένων. Παράδειγμα, πρόσβαση στους ελέγχους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να μην έχουν πρόσβαση όλοι στις πληροφορίες γιατί υπάρχουν και εμπορικά συμφέροντα εδώ. Το ηλεκτρονικό κομμάτι, ναι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν ξέρω ποια γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί, XML ή κάτι άλλο Πάντως ίσως θα μπορούσαμε στο παράρτημα της οδηγίας να έχουμε τη δυνατότητα Διακόπτει ο Πρόεδρος, υπάρχει πρόβλημα με τη διερμηνία γιατί έχουμε θόρυβο στα μεγάφων για τους διερμηνείς. Υπάρχει πρόβλημα και με τον αέρα εδώ πέρα. Είναι πολύ άσχημος ο αέρας, πρέπει να ανοίξουμε και ένα παράθυρο εδώ μέσα. Is it better now? Okay. So Ωραία. Σταμάτησε ο θόρυβος. Εντάξει, ο θόρυβος για τον αέρα θα πρέπει να το εξετάσουμε. Λοιπόν, για τα τελευταία αυτά σημεία. Ένα, πρόσβαση σε ελέγχους. Σημαντικό. Δεύτερον, η ηλεκτρονική μορφή και μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί ίσως θα έπρεπε να μπει στα παραρτήματα όχι στο διατακτικό της οδηγίας για να μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα αλλαγές. Όσον αφορά τις εσωτερικές μεταφορές, μου φαίνεται ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί το έχουμε προσπαθήσει και οι δυνατότητες interoperability μεταξύ εσωτερικών πλωτών μεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών υπάρχουν. Για παράδειγμα, όταν ε, ξεκινάμε τη μεταφορά με θαλάσσια μεταφορά και περνάμε στη συνέχεια στις εσωτερικές μεταφορές, το θέμα των γλωσσών. Όντως, όταν μιλάμε για θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να πούμε ότι ουσιαστικά τα αγγλικά είναι η κοινή γλώσσα που χρησιμοποιείται. Γιατί σε κάθε πλοίο υπάρχουν ναυτικοί από διάφορες γλώσσες. Τώρα το τι είδου αγγλικά μιλάμε μπορεί να είναι μισά αγγλικά, μισά φιλελεπινέζικα. Όμως καταφέρνουν να συνεννοούνται και τουλάχιστον διευκολύνονται οι επικοινωνίες στους λιμένες με τους πιλότους κτλ. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρεται και η χρήση κοινή γλώσσα σε διάφορες συμφωνίες. Είναι θέμα ασφάλειας. Επί της αρχής Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι συμφωνούμε με την έκθεση, είναι πολύ καλή έκθεση και θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία πολύ σύντομα με το Συμβούλιο. Να πω εδώ ότι βελτίωσε το κείμενό μας το Συμβούλιο, πρέπει να είμαι ειλικρινής εδώ, μας βοήθησαν και υπάρχουν πράγματα που συμπεριλήφθηκαν από το Συμβούλιο που αναφέρει και ο εισηγητής σας άρα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε τους επόμενους μήνες προκειμένου ή δυνατόν να καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Γιατί νομίζω ότι όλοι επιθυμούμε να επιληθεί αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις θαλάσσιες μεταφορές. Τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα. Τελωνία, υγειονομικές διαδικασίες, στο μέλλον ε, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση ενδεχομένως με χρήση του Γκαλιλαίου, κάτι που θα διευκολύνει πολύ τα πράγματα όσον αφορά τον εντοπισμό των ε, φορτίων όλα αυτά βεβαίως για το δεύτερο μισό της δεκαετίας που θα έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε όλους για την πολύ χρήσιμη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ. Κύριε Στέρξ, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση που ήταν χρήσιμη και πολύ θετική για το έργο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους για τα καλά τους λόγια και τον ε, συνάλφο της ε, Κομισιόν γιατί είχαμε ήδη ανταλλάξει απόψεις ε, τους περασμένους μήνες. Αναμένω και τις τροπολογίες, βελτιώσεις των συναδέλφων όπου επιδέχεται βελτίωση οπωσδήποτε θα το κάνουμε. Τώρα να αναφερθώ σε κάποια ερωτήματα που ε, οι τεχνικές προδιαγραφές, μήπως είναι πάρα πολύ ε, περιοριστικές. Ε, μην νομίζετε πως εγώ τα ξέρω όλα. Εμένα μου είπαν οι άνθρωποι που ασχολούνται στην πράξη ναι, Πώ έτσι πρέπει να το διατυπώσετε για να είναι σαφέ το τι πρέπει να συμβεί, αλλά να είναι αρκετά ευρύ. Αν δεν ισχύει αυτό, υποθέτω πω από αύριο θα αρχίσουν να έρχονται τα email από του ειδικού που θα μου πούνε όχι, δεν πρέπει να λέτε TMX αλλά TMA κτλ. Θα το δούμε αυτό. Συνήθω γρήγορα ε, οι άνθρωποι αντιδρούν πράγματι και λένε ότι δεν πρέπει να κάνετε αυτό αλλά το άλλο. Οπότε θα ακούσω τι, τι θα πούν οι ειδικοί όσον αφορά τη γλώσσα. Νομίζω πως ε, εντός του IMO ούτως ή άλλως ε, στις ε, συμβάσεις περί ασφάλειας όπως η Σόλας παραδείγματος χάρη λένε πως στο πλοίο και στην επικοινωνία μεταξύ πλοίου και ξηράς ακτής ε, ε, για ασφάλεια. Όπως είπε και ο κύριος Φαντάλη ακόμα και στην εσωτερική ναυσιπλοεία έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι από πιο εξωτικές χώρες, ας τις πούμε έτσι. Οπότε για την ασφάλεια είναι απαραίτητο να υπάρχει κατανόηση. Και στην περίπτωση αυτή νομίζω πως ε, και η επικοινωνία δεν πρέπει να είναι τόσο δύσκολη. Δεν θα με συζητήσουν τώρα φιλοσοφικά δοκίμια εδώ πέρα. Πέντε πρακτικές πληροφορίες να συνεννοηθούν και πρέπει να ξέρουν αυτούς τους πέντε όρους. Και ε, μπορούμε, ξέρω εγώ, να το γράψουμε το, νούμερο ένα ότι είναι αυτό και στα βουλγαρικά και στα ολλανδικά και στα οτιδήποτε. Και δεν μιλάμε βέβαια για να μιλάει κανείς απτέστος ε, τη γλώσσα, απλά για να υπάρχει μία σύμβαση να μπορούν να συνεννοηθούν. Ρωτήσατε, κύριε Φώστερ, τι γίνεται αν υπάρχουν φορτία σε ένα κοντέινερ για εντός και εκτός της Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θα ανοίξουν το κοντέινερ στο λιμάνι και θα χωρίσουν το φορτίο. Αλλά εγώ δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Ε, συνήθως μένει κλειστό μέχρι το τελικό του προορισμό το κοντέινερ. Για την απίθανη περίπτωση πρέπει να ανοίξει ένα κοντέινερ μέσα στο λιμάνι, νομίζω πως ε, πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα. Αλλά είναι περιπτώσεις νομίζω που μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού γιατί συνήθως παραμένουν κλειστά και πάνε μετά σε ένα κέντρο logistics και δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το οποίο λέτε για τα μικρά λιμάνια και την ευελιξία. Θα το δούμε αυτό, ίσως να καταθέσετε κάποια τροπολογία, αλλά πρέπει να προσέξουμε η επένδυση που απαιτείται από ένα λιμάνι δεν είναι τεράστια να έχει ένα PC και ένα προγραμματάκι. Ε, μπαίνει αμέσω ε, στο σύστημα. Δεν είναι καμία τεράστια επένδυση κέντρο πληροφορικής, είναι κάτι το απλό. Αλλά αν υπάρχουν λιμάνια που έχουν προβλήματα, μπορούμε να το δούμε αυτό με την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα πόσα είναι αυτά τα προβλήματα και δεύτερον πώς θα λυθούν ε, με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά εντάξει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα μικρά λιμάνια αλλά μετά πόσο ορίζει στα μικρά λιμάνια. Τόσο θα το δω έτσι με θετικό πνεύμα. Καταθέστε και μία τροπολογία. πρέπει να προσέξουμε όμως. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κούν Μιλάω, ρωτήστε για το IES. Το IES είναι ένα σύστημα το οποίο ισχύει για την ε, κυκλοφορία, για την κίνηση και αν υπάρχει επικίνδυνο φορτίο. Μιλάει δηλαδή για επικίνδυνα αγαθά. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για όλα τα δεδομένα του φορτίου. Και δεν λέμε μόνο τι είναι κίνδυνος για την αυτιλία, αλλά τι ε, ε, μπαίνει και τι βγαίνει. Οπότε είναι πολύ ευρύτερο το, το αντικείμενο. Μπορεί για ένα πλοίο με κοντέινερ να έχουμε ένα ε, σύντομο μήνυμα του στο ΑΕΣ που να λέει δεν έχουμε επικίνδυνο φορτίο, αλλά εάν έχει 5.000 κοντέινερ χωρίς κανένα επικίνδυνο φορτίο, σε αυτό το σύστημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα. Με το τι υπάρχει δηλαδή μέσα σε αυτά τα 5.000 κοντέινερ. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει... Ε, επικάλυψη και διπλή χρήση και των δύο συστημάτων, αλλά θα μπορούσαν όλα αυτά τα δεδομένα να περνάνε μέσω του SafeSynet, να, να υπάρχουν όντω, αλλά να μην δίνονται δύο φορές τα ίδια στοιχεία. Αλλά αυτό νομίζω θα τα αφήσουμε στα χέρια των ειδικών. Αλλά εκεί νομίζω μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντω το Γαλιλαίο όσον αφορά π.χ. την παρακολούθηση και ταυτοποίηση των κοντέινερ. Αν μπορεί να γίνει αυτό ηλεκτρονικά, θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα, πάρα εύκολα και τα, τα έγγραφα. Δηλαδή μια λίστα ποια θα μείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια ε, πάνε σε τρίτες χώρες ή έρχονται από τρίτες χώρες και αν μπορούμε αυτά να τα ταυτοποιήσουμε και ηλεκτρονικά γίνεται και πολύ πιο εύκολη η δουλειά μας, αλλά αυτό προσεχώς όταν θα έχουν ξεκινήσει τα πράγματα και θα έχει υπάρξει μία επένδυση αλλά οπωσδήποτε θα γίνονται δύο διαφορετικοί λίστες για το φορτίο, για το τι είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι είναι εκτός και όταν θα χρησιμοποιούμε το Γαλιλαίο. Τώρα για τους πιλότους φλεγούς. Ενδιαφέρον είναι να δούμε. Πως δεν μιλάμε για κινδύνους που θα διατρέξουμε εδώ πέρα. Είναι προφανές πως ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια ή όποιος ε, ασχολείται με τους πλοηγούς μπορεί να περάσει ένα κανόνα και να λέει εδώ είναι υποχρεωτικός ο πλοηγός όπως π.χ. ένα κομμάτι στη Βαλτική μεταξύ Βαλτικής και Βόρειας θάλασσας είναι υποχρεωτικός ο πλοηγός. Εγώ δεν λέω πως πρέπει να καταργηθεί εκεί πέρα. Απλά σε κάποια κράτη-μέλη το ε, πιστοποιητικό αυτό γίνεται τόσο δύσκολο ώστε θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο απλή ε, ναυτιλία αν θέλετε ε, αν ξέραμε ποια είναι τα, τα κριτήρια. Έχω παράδειγμα, έχω ακούσει για καπετάνιους που σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάνουν ένα δρομολόγιο, μετά πάνε σε άλλο δρομολόγιο, αλλά δεν μπορούν να διατηρήσουν το πιστοποιητικό τους γιατί πρέπει να πηγαίνουν στο ίδιο λιμάνι ε, χύψη φορές εντός του ίδιου μήνα και μετά χάνουν το πιστοποιητικό. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Δηλαδή δεν α, ε, τους δίνουν τα, τα πιστοποιητικά. Ενώ κάποιο τέτοιο μέτρο να προστατεύσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Οπωσδήποτε Νομίζω πως υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία εδώ εντός αίθουσας. Αλλά μετά θα γίνει και η συζήτηση με το, με το Συμβούλιο. Ε, όσον αφορά την ημερομηνία, είναι δύσκολο πράγματι εντός του Συμβουλίου και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε Συμβούλιο πως δεν μπορούμε να περιμένουμε γιατί είναι επίγοντο ζήτημα. Γνωρίζω επίσης πως συζητάνε στο Συμβούλιο να μην ισχύσει αυτή η οδηγία στα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ακτογραμμή, αλλά πρέπει να ισχύσει για τα κράτη-μέλη που έχουν σημαία. Μπορεί να μην έχουν ακτή, αλλά να έχουν σημαία. Και να υψώνουν δηλαδή τα πλοία τη σημαία τους. Πρέπει και αυτοί να εφαρμόσουν την οδηγία. Είναι μια δύσκολη συζήτηση στο Συμβούλιο αλλά νομίζω πως ε, δεν το συζητάμε εδώ πέρα ε, στο Κοινοβούλιο λεωτούμε. Επίσης αναμένω κάποια συζήτηση για τη γλώσσα και για τους ε, πλοηγούς. Νομίζω πως εκεί θα μας προξενήσει δυσκολίες το Συμβούλιο, αλλά εγώ το βρήκα εντό τη ανακοίνωση. όπου είναι στα, στα μακροπρόθεσμα για το τι θα γίνει με το πακέτο των λιμένων αναφέρονται και οι πλοηγοί εκεί πέρα Οπότε πρέπει νομίζω να πούμε κάτι να ξεκινήσει συζήτηση με το Συμβούλιο. Και ελπίζω συνάδελφοι να τελειώσουμε το συντομότερο το δυνατόν για να ξέρουν και τα λιμάνια και τα κρατημέλη ποιο είναι το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και αναμένω και μια καλή συζήτηση με το Συμβούλιο που είναι πάντα ευχάριστη και βεβαίως και εμείς θα συνεισφέρουμε στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέρξα. Να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα για αυτή την έκθεση. Προβλέπει προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών στις 27 Φεβρουαρίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 22 Μαρτίου. Η υιοθέτηση στην Επιτροπή στις 23 Μαρτίου. Ενώ η συζήτηση στην Ολομέλεια προβλέπεται μεταξύ του Απριλίου και του Μαΐου του 2010. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. <clears throat> Σχέδιο γνωμοδότηση για την απαλλαγή της Επιτροπής, η κυρία Γιάλα Σεντέρ έχει ήδη έρθει. Είναι έτοιμη προς διαπραγμάτευση. Κυρία Γιάλα Σάντες, Έχετε το λόγο για την απαλλαγή 2008. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ζητώ συγγνώμη αν δεν πρόσεχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή στην Επιτροπή Μεταφορών παρεμβαίνω με δύο ιδιότητες, γιατί βεβαίως είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει, αλλά και γιατί ε, είμαι μέλος και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Η δυνατότητα λοιπόν που μου δόθηκε να κάνω αυτή την έκθεση για την ε, απαλλαγή είναι κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τη σύντομη αυτή γνωμοδότηση, θα προσπαθήσω, <clears throat> αφού κάνω μία ανακεφαλαίωση των γεγονότων, να, σημίσω, να μιλήσω για ορισμένους φορείς, όχι τους εκτελογικούς, που σε ό,τι αφορά τη ευρωπαϊκά δίκτυα αποτελούν το θέμα της έκθεσής μου, θα ήθελα όμω να εντοπίσω ορισμένα σημεία, ορισμένε πτυχέ που επαναλαμβάνονται για το λόγο αυτό ζητάμε περισσότερες εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο ε, επανέρχονται ορισμένα κονδύλια ιδιαίτερα ε, ευαίσθητα όπως η ασφάλεια των μεταφορών, τα δικαιώματα των επιβατών. Είναι αλήθεια σιγά σιγά αρχίζουν τα πράγματα να καλυτερεύουν. Σε κάθε περίπτωση όμως μας εντυπωσιάζει ότι οι πιστώσεις πληρωμών έχουν ε, χρησιμοποιηθεί μόνο κατά το 27%. Πάρα πολύ ε, μεγάλο ποσοστό απορρόφησης. Η Επιτροπή ελπίζω να μπορέσει να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Λαμβάνω υπόψη το γεγονός ότι το ελεκτικό συνέδριο κάνοντας μία αντιπαράθεση μεταξύ της πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης και της Επιτροπής Μεταφορών επικεντρώθηκε περισσότερο στην πρώτη. Γιατί αν κάνουμε μία σύγκριση, η πολιτική μεταφορών δεν κερδίζει και πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα κονδύλια αυτά. Γι' αυτό ακριβώ στο σημείο 3 αναφέρω ότι το Κοινοβούλιο επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη χρηματοδότηση των δικτύων. Θα ήθελα όμως να θυμίσω στις χώρες μέλη ότι θα πρέπει και εκείνα με τη σειρά, εκείνες με τη σειρά τους να συμβάλλουν. Θα πρέπει να το κάνουμε όπως γίνεται με τα διερθωτικά κονδύλια. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτά τα προγράμματα των διευρωπαϊκών δικτύων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο, είναι ένα άλλο ανησυχητικό θέμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε από κοντά στην Επιτροπή αυτή. Όχι μόνο το ξεκίνημα, του προγράμματος ε, Γκαλιλαίου αυτού καθ' αυτού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόζεται ο προπολογισμό. Μιλάμε, γενικά υπάρχει κακή άποψη για τον Γαλιλαίο και γι' αυτό το λόγο είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Είναι, υπήρξε μια υποαπορρόφηση των πιστώσεων, υπήρξε μια κρίση, ξεκίνησε μια καινούργια περίοδο. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μα δώσει ορισμένε εξηγήσει και αυτό ελπίζω να γίνει σε λίγο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι παρόλο που υπάρχει ένας δείκτης λάθους που για τα άλλα κονδύλια είναι υψηλότερο παρατηρείται μία πτωτική τάση μολονότι σε ό,τι αφορά μία πολιτική εσωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που πρόκειται για προγράμματα που δεν θα πρέπει να συνεπάγονται τόσες δυσκολίες ή τόσα λάθη μετά από τόσο καιρό. Με χαροποιεί το γεγονός ότι τα, οι διάφοροι λογαριασμοί του εκτελεστικού φορέα με ικανοποιεί όπως έλεγα το γεγονός ότι οι λογαριασμοί αυτοί θεωρούνται απόλυτα ε, κανονικοί. Είναι αλήθεια ότι με αργούς ρυθμούς γίνεται πρόσληψη του προσωπικού ίσως με πολύ αργούς ρυθμούς, το είπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λογικό να υπάρχουν καθυστερήσει. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ναι στην απαλλαγή για το κεφάλαιο που αφορά τις μεταφορές στην Επιτροπή. Παρόλα αυτά, πριν γίνει αυτό, θα επιθυμούσα να ακούσω τις εξηγήσει, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που ανακύπτουν συνέχεια, όπως για παράδειγμα η απορρόφηση των ε, ε, πιστώσεων πληρωμών για το Μάρκο Πόλο. Θα πρέπει να ακούσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αποφασίσουμε. Παραμένω στη διάθεσή σας ε, είμαι απόλυτα ανοιχτή σε σχόλια και σε τροπολογίες που θα υποβληθούν από τους συναδέλφους. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά την περίοδο υποβολής των τροπολογιών, το μέρος εκείνο που αφορά τον τουρισμό δεν ελήφθη υπόψη μέχρι στιγμή από την Επιτροπή. Και ύστερα υπάρχει το πρόβλημα της υποαπορρόφησης των πιστώσεων που δεν αναφέρθηκε και που είπα ότι θα τροποποιηθεί, αλλά δυστυχώς δεν είχα το χρόνο να το εντάξω σε αυτή την ε, γνωμοδότηση. Σε κάθε περίπτωση είμαι ανοιχτή στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρός, παρακαλώ, για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να αναφερθούμε στη συζήτηση που ξεκίνησε χθε με τους διάφορους φορείς. Μία απαλλαγή θα πρέπει να έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Συγγνώμη, πάλι έχουμε πρόβλημα με τα μικρόφωνα και τη διερμηνία. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Monsieur vous pouvez continuer.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 η συζήτηση για την απαλλαγή θα έπρεπε να είναι και πολιτική συζήτηση. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε όλοι παρόμοιες διαπιστώσει. Είναι αλήθεια ότι συχνά όταν συζητείται ο προϋπολογισμός αυτό που ζητάμε κυρίως ήταν, είναι αύξηση των κονδυλίων Ίσως λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να μιλήσουμε για σημαντικούς τομείς. Για παράδειγμα, το Μάρκο Πόλο είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και εκεί έχουμε απορρόφηση κατά 40%. Γιατί είναι τόσο χαμηλό αυτό το ποσοστό ή τι είδους προτάσεις μπορούμε να κάνουμε εδώ. Μήπως πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια στο Μαρκοπόλε. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει και στο παρελθόν, αλλά το να κάνουμε απλά κάθε χρόνο την ίδια διαπίστωση δεν βοηθάει. Το ίδιο ισχύει και για το Γαλιλαίο ίσως δεν επαρκούν τελικά τα κονδύλια. Μπορεί να μην μπορούμε να εξετάσουμε όλον τον προϋπολογισμό, αλλά ίσως θα έπρεπε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα δείγματα, αυτό το 2-5% για τους ελέγχους. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά κονδύλια τα οποία εγκρίνονται αλλά τελικά δεν χρησιμοποιούνται στη διάρκεια του έτους. Οπότε μήπως αυτές τις γραμμές θα έπρεπε να τις επανεξετάσουμε, για παράδειγμα στο Μαρκοπόλο. Μήπως θα έπρεπε να μεταφέρουμε κονδύλια στα διευρωπαϊκά δίκτυα όπου συνήθως είμαστε στο περίπου 100% της απορρόφησης. Εν πάση περιπτώσει σίγουρα ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς και ενδιαφέρουσα θα είναι η συζήτηση. Ευχαριστώ. Το λόγο στον κύριο Κραμέρ. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την εισαγωγή της. Όντως, μας θυμίζει το παρελθόν αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν όμως κάποιες παρατηρήσεις που είναι σωστές και πάλι όντες θα έπρεπε να κάνουμε μία συζήτηση και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κονδύλια για τις μεταφορές. Βλέπουμε σε ορισμένες περιπτώσεις απορρόφηση 27%. Βλέπουμε περιπτώσεις όπου ναι μεν θεωρείται δεδομένο ότι θα μπορεί κανείς να αγοράσει βινιέτες σε όλη την Ευρώπη αλλά θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιες χώρες της Ευρώπης έχει εφαρμοστεί όντως αυτό. η Υπουργό κ. Τσιπρίσα ε, το παρουσίασε να ήταν δική της ιδέα. Όμως, τελικά, τι συμβαίνει εδώ. Και αν δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αυτή η πολιτική, τι πρέπει να κάνουμε για να εφαρμοστεί. Πριν από δύο-τρία χρόνια είχα κάνει κι εγώ εισηγητής για αυτή την έκθεση το 2007 και τότε στο σημείο 7 ζητούσαμε από την Κομισιόν να μας ενημερώνει κάθε χρόνο με λεπτομερή έκθεση για τα προγράμματά της. Αλλά ούτε και τώρα βλέπουμε κάτι τέτοιο. Πού βρίσκονται αυτές οι εκθέσεις. Μπορούμε να τις εξετάσουμε. Υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις. Είχαμε συμφωνήσει επ' αυτού του θέματος με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά τελικά και τώρα σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε πάλι δεν βλέπουμε αυτές τις εκθέσεις. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω με τους ε, προλαλήσατες για ορισμένα θέματα. Καταρχάς ευχαριστούμε την κυρία Γιάλα Σεντερ για την έκθεσή της. Όντως ε, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής στη διάρκεια του έτους, αλλά θεωρώ ότι για παράδειγμα εδώ στο σημείο 7 ζητάτε από την Κομισιόν περισσότερες διευκρινήσεις Πώς μπορείτε να εξελογήσετε την ελληπή εξελόγηση και τι, την ελληπή απορρόφηση και τι μπορείτε να κάνετε για να την ε, προωθήσετε έτσι ώστε αυτά τα οποία είναι προϋπολογισμένα για τις μεταφορές να χρησιμοποιούνται και κατά τα λοιπά συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ αν ε, εξαντλήσουμε το 27% των μέσων μόνων δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό και το γεγονός ότι παραδείγματο χάρη η Ευρώπη θα μπορούσε να βρει μια άλλη λύση όσον αφορά τα ειστήρια. Το συζητήσαμε άμεσα και με τον κύριο Επίτροπο. Δεν αφορά καθόλου τα... το κόστος. Νομίζω αξίζει και αυτό να το αναφέρουμε. Επίσης το ποστό σφάλματος και αυτό δεν είναι μεταξύ 2 και 5%. Πρέπει να είναι χαμηλότερο. Αλλά το βασικό το είναι αυτό που είπαν και οι προλαλήσαντες. Ε, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να απορροφηθούν πράγματι αυτά τα μέσα και πράγματι έχει δίκιο ο κύριος ε, γκρος μπορούν να αφιερωθούν σε κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι του προπολογισμού, αλλά πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Γνωρίζουμε γενικά πόσο σημαντικό είναι το μέσο μεταφορών για την εσωτερική αγορά. Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρούτσι από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να απαντήσω γενικά επί του συνόλου. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι πιστώσεις ανάληψη ε, υποχρεώσεων είναι διαφορετικές από τις πιστώσεις πληρώμου. Μπορούν να γίνουν οι πληρωμές μόνο με τιμολόγιο, με επίδειξη τιμολογίου ή κατόπιν ετήσεω. Σε ό,τι αφορά τα τρία σημεία, το, την ασφάλεια των μεταφορών, τα δικαιώματα των επιβατών και το Μάρκο Πόλο, πιστεύω ότι θα μπορούσα να πω ότι το πιο σημαντικό, το Μάρκο Πόλο, το οποίο αφορά σημαντικά κονδύλια, αποτέλεσε αντικείμενο μίας επανεξέτασης και το ποσοστό εκτέλεσης το 2009 ήταν γύρω στο 100%. Φτάσαμε στο σημείο να ενισχύσουμε το κονδύλιο με άλλες ε, πληρωμές λόγω της επιτυχίας του Μάρκο Πόλο. Συνεπώς η αναθεώρηση επέτρεψε να επιτύχουμε μια εξισορρόπηση με την κακή εκτέλεση του 2008 σαν αποτέλεσμα των επιλογών που έγιναν. Μερικές φορές λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τεχνικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Γκαλιλαίο, πιστεύω ότι θα μπορούσα να πω ότι το 2008 ήταν μια μεταβατική χρονιά η οποία χρησιμοποιήθηκε βασικά για να ε, επιτευχθεί συμφωνία των αντιπροσωπιών με την European Space Agency και τη μεταφορά του προσωπικού. Το προσωπικό αυτό έφτασε στο τέλος του 2008. Το 2008 υπογράψαμε τη συμφωνία και το 2009 όλες οι συμβάσεις, το μεγαλύτερο μέρος των ε, συμβάσεων αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το 2008, μεταβατική χρονιά, το 2009 ξεκίνησε η συνήθιες διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την ε, ΤΕΝΤΕ, δηλαδή σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το προσωπικό, Μπορώ να σας πω ότι έχει ένα ελάχιστο επίπεδο κενών θέσεων. Μόνο δύο κενές θέσεις, θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί. Και μιλάμε για 100 άτομα περίπου προσωπικό. Μιλάμε για ένα ποσοστό φυσιολογικό. Το 2008 δεν έγιναν πολλές προσλήψεις. Το 2008 ήταν η χρονιά μετά από την απόκτηση αυτονομίας από τον ε, φορέα. Μετά τα πράγματα άρχισαν να πήραν το φυσιολογικό του ρυθμό και μερικές φορές χρειάζονται 4, 5, 6 μήνες μέχρι που να επιτευχθεί αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση του κυρίου Κράμερ, γιατί δηλαδή αυτό το 27% της εκτέλεσης για τα δικαιώματα των επιβατών είναι κάτι ανησυχητικό ή όχι. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι σε ό,τι φορά το κεφάλαιο δικαιώματα επιβατών, το κονδύλιο ήταν 350.000 ευρώ. Το κοινοβούλιο, τη μεγάλη του σοφία, το έφτασε στα 750.000. Εμείς θα έπρεπε να εξετάσουμε διάφορες εφαρμογές αυτής της στρατηγικής. Πιστεύω ότι έδωσα το λόγο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Φιλίπ, θα σας δώσει τις λεπτομέρειες που θα θέλατε να ακούσετε. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο κύριος Μπανούτσι, το 2008 Είχαμε επιπτώσει ανάληψη υποχρεώσεων για αυτό το κονδύλιο και δύο δραστηριότητε που προβλέπονται. Ήταν μια ενημερωτική εκστρατεία για τα δικαιώματα των επιβατών και μια διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Η δεύτερη δραστηριότητα είναι εκείνη που έλαβε χώρα και ενώ αποφασίστηκε να αναβληθεί η πρώτη εν των προτάσεων που δεν είχαν ακόμα υποβληθεί. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε τώρα είναι ότι επίκειται ε, μία εκστρατεία, ένα project για να αξιολογήσουμε τι βελτιώθηκε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών αλλά και για να υπάρξει μεγαλύτερη ε, ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών και για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες που προετοιμάζονται και που αφορούν τις θαλάσσιες και χεσές μεταφορές. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που μας απασχολεί για φέτος. μετά από τα όσα εφαρμόστηκαν το 2008. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Βανούτσι σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών. Η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει 350.000 ευρώ για πιστώσεις πληρωμών. Μας δόθηκαν 728 δαπανήθηκαν 200.000. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μικρότερο ποσό από αυτό που ζητήσαμε. Είναι γύρω στο 55%. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. Michael, το, δικό μου το ερώτημα για τις εκθέσεις που πρέπει να μας κάνετε κάθε χρόνο. Δεν έχω ξαναδεί η παρέμβαση της Κομισιόν να προκαλεί τόσο πολλές αντιδράσεις ταυτόχρονα και για τόσα πολλά θέματα. Οπότε να σας ακούσουμε πρώτα εσάς, μετά Ματίας, Σινές και μετά η συγγήτρια. Μάικλ, ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ναι, μα την είχα θέσει. Η έκθεσή μου της 1ης ε, Τρίτου 2007 την έχετε νομίζω. Παράγραφος 7 προτείνει κάθε χρόνο να έχουμε μια λεπτομερή έκθεση. Και ρώτησα πού μπορούμε να την, να την βρούμε ή εάν δεν υπάρχει. Αυτό ήταν όλο. Να τα πω στα γαλλικά μήπως ε, είναι καλύτερα ποιο είναι το ποσοστό δειγματοληψίας για όλες ε, τις ε, περιπτώσεις. Ε, μιλάτε για διακύμανση μεταξύ 2 και 5% μήπως έπρεπε να είναι 5 ως 10%. Και το δεύτερο θέμα, ακόμη πιο σημαντικό, υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης ορισμένων γραμμών που χρησιμοποιούνται σχεδόν κατά 100% τα κονδύλια. Μήπως μπορούμε, αν περισσεύουν χρήματα από αλλού, να ενισχύσουμε αυτές τις γραμμές. Γιατί πάντα προσπαθούμε να ενισχύσουμε λίγο τα κονδύλια για αυτές τις γραμμές. Και εγώ προσωπικά λυπάμαι εφόσον ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση των μεταφορών, να μην μπορούμε να ενισχύσουμε κάποιες γραμμές όπου υπάρχει απορρόφηση σχεδόν 100% τουλάχιστον για τις πιστώσεις πληρωμών αυτό. Περιμένω την απάντησή σας ειδικά για το δεύτερο θέμα. Κύριε Σέντερ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπονούτσι για τις πληροφορίες. Όμως, μία ερώτηση για τον Καλλιλέο. Ναι, υπάρχει θέμα με τη μεταφορά του προσωπικού κτλ. Όμως αυτή τη στιγμή ως ποσοστό των πιστώσεων ε, πληρωμών θα υπάρξει βελτίωση πάνω από αυτό το 50%. Κύριε Μπονούτσι, τρία επιπλέον ερωτήματα προφανώς επειδή θεωρούν ότι δεν απαντήσατε την πρώτη φορά. Ναι, γιατί είχαν γίνει πολλές ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω με τον Γαλιλαίο. Θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση πώς. Η απάντηση είναι απλή. Για το 2009 βρισκόμαστε στο 100%. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να σας καλύψει τον Γαλιλαίο μπορεί να αντιμετωπίσει όλα άλλα προβλήματα, αλλά όχι προβλήματα υλοποίησης. Μέχρι στιγμής έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα για το 2009. Όσον αφορά τώρα το ποσοστό σφάλματος που ανέφερε ο κύριος Γκρός, κοιτάξτε, το μέγεθος του δείγματος αποφασίζεται από το ελεγκτικό συνέδριο. Συνήθως είναι πολύ μικρό. Να σας πω, αν θέλετε, τι κάνουμε εμείς τους ελέγχους μας, αν σας ενδιαφέρει. Συνήθως ελέγχουμε την πιο σημαντική σύμβαση από άποψη μεγέθους κονδυλίων. Μετά Χρησιμοποιούμε ένα τυχαίο δείγμα για ελέγχους και επιπλέον ορισμένα δείγματα των συμβάσεων που θεωρούμε ότι είναι οι πιο επικίνδυνες με βάση τις εμπειρίες μας στο παρελθόν. Αυτή είναι η μέθοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης κάνουμε και προληπτικούς ελέγχους προκειμένου να ενημερώνουμε τους δικαιούχους για το πώς μπορούν να συμμορφωθούν. Και επιπλέον κατά τη διάρκεια της σύμβασης, γιατί προσπαθούμε πάντα να προλαμβάνουμε τα προβλήματα, Οργανώνουμε λοιπόν σεμινάρια με τους δικαιούχους προκειμένου να είναι σαφές το τι προβλέπεται από τις συμβάσεις τους και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε το ποσοστό σφαλμάτων που συνήθως προκύπτει. Άλλα ερωτήματα? Για τις μεταφορές. Στην καθημερινή μας ζωή όντως ζητάμε συχνά μεταφορές για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. όταν θεωρούμε ότι κάποιες πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλη γραμμή του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, το 2008 είχαμε κάτι κάτω από το 98% χρήση των πιστώσεων δεσμεύσεων ανάληψη υποχρεώσεων. Βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Κρόσ, υπάρχει κάποια διαφορά όταν μιλάμε για πιστώσει πληρωμών, γιατί εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι δικαιούχοι. Εν πάση περιπτώσει, περίπου τον Οκτώβριο κάθε χρόνο έχουμε κάποιες συνολικές μεταφορές, όπως τις αποκαλούμε. Πάντως, ακόμη και με αυτές τις διαδικασίες δεν είναι τα πράγματα τέλεια, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι πρόκειται να γίνει, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά ποσά για την τον τελευταίο καταμερισμό των χρημάτων. Να απαντήσω και στον κύριο Κράμερ για τις εκθέσεις. Προφανώς υπάρχει κάποια παρανόηση εδώ. Εμείς κάνουμε έκθεση στη γάμα δέλτα προϋπολογισμών για κάθε μια γραμμή και η γάμα δέλτα προϋπολογισμών είναι αυτή η οποία πρέπει να δώσει εκθέσεις σε εσάς. Ίσως λοιπόν πρέπει να αποκτήσετε απευθείας επαφές με τη γάμα δέλτα προϋπολογισμών. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να σας διαβιβάζουμε εκθέσεις για την εφαρμογή των προϋπολογισμών τόσο για τις, πληρωμές, για τις πιστώσεις πληρωμών όσο και για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Πρόεδρος, υπάρχουν κάποια επικίνδυνα θέματα εδώ. Αυτό που λέει ο κύριος Κράμερ είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τις ετήσιες εκθέσεις, αλλά δεν τις έχουμε λάβει. Σημειώστε όμως, παρακαλώ, ότι η έκθεση για ένα έτος οριστικοποιείται τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Άρα για το 2009 η έκθεση θα είναι έτοιμη τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου. Αν θέλετε μπορούμε να σας τη διαβιβάσουμε. Ναι, αυτό θα θέλαμε. Κυρία Αγιά Λασαντέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα μιλάμε για την απαλλαγή του 2008. Συνεπώς οι εκθέσεις, όπως είπε η κυρία Γράμμε, θα έπρεπε να μας έχουν δοθεί πέρσι. Σε κάθε περίπτωση θα ήμασταν ευγνώμονε στην Επιτροπή εάν θα μπορούσε να μα στείλει ένα αντίγραφο αυτών των εκθέσεων, κυρίω γιατί τα πολιτικά προγράμματα που μερικέ φορέ με κόπο εντάσσουμε στον προπολογισμό, θα πρέπει να δίνονται μάχες με την Επιτροπή Προπολογισμών έχουν ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο ε, εκτέλεση, απορρόφησης ε, και η εικόνα που δημιουργείται δεν είναι και τόσο καλή. Δυστυχώ ο συνάδελφο έφυγε. Θα ήθελα να επιμείνω και να μου παραθέσουν οι συναδελφοί τα παραδείγματα που αφορούν το ελεγκτικό συνέδριο και τις επαληθεύσεις που κάνει. Αυτό είναι ένα πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό. Με τον πρόεδρο κύριο Καλτέρα είπαμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια πιο διαφανή κατάσταση. Πρόκειται για μια εσωτερική ε, αναθεώρηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα στοιχεία επικινδυνότητας ε, για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και σε ό,τι αφορά το θέμα της εκτέλεσης. Σε ορισμένους τομείς υπήρξαν έγιναν βελτιώσει, Μόνο ότι μιλάμε για τα ποσά, για τα κονδύλια του 2008. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και περιμένω περαιτέρω σχόλια. Η προθεσμία 3η Φεβρουαρίου, 27 θα συζητηθούν οι τροπολογίες και η ψηφοφορία θα γίνει 28 Φεβρουαρίου και πιστεύουμε ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα ψηφίσει στις 3 Μαρτίου. 27 λοιπόν θα συζητηθεί η ψηφοφορία 28. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο διάλειμμα πριν καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας Κάντε μου τη χάρη να επιστρέψετε στις 11 και αυτό το διάλειμμα θα δώσει τη δυνατότητα στην Ισπανική τηλεόραση να εγκαταστήσει τα μηχανήματά της χωρίς να μας ενοχλήσει. Ελπίζω να έρθετε ε, καλοντημένοι γιατί σε 15 λεπτά θα σας πάρει η Ισπανική τηλεόραση. Διακόπτουμε μέχρι τις 11. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνάδελφοι. Can I welcome to... Καλώς ορίζω στην Επιτροπή την Πρόεδρεους τον Προεδρεύοντα τον κύριο Μπλάνκο Λόπες τον κύριο Υπουργό λοιπόν. Οι συνάδελφοι εδώ πέρα αναμένουν με αγωνία το τι έχετε να μας πείτε για την Ισπανική Προεδρία και οπωσδήποτε αν το παρελθόν μας διδάσκει τίποτα τότε θα έχουν και ερωτήσεις, ίσως και δύσκολες ερωτήσεις για να απαντήσετε στο χρόνο που μας απομένει. Ε, Σήμερα χτυπάμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Έχουμε εσάς εδώ το πρωί και έτσι για να συνέλθουμε λίγο έχουμε τον συνάδελφό σας του τουρισμού το απόγευμα. Οπότε αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στην Ισπανική Προεδρία και στο τι μας προτείνεται. Ξέρω πως έχετε ξαναέρθει και πριν ξεκινήσει η Ισπανική Προεδρία, κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο για εμάς. Χτες ε, η Σουηδέζα υπουργό τελείωσε, ολοκλήρωσε την δική της Προεδρία και λογικό είναι την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε με εσάς. τον νέο Προεδρεύοντα. Και Αναμένουμε την συνεργασία μαζί σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Οπότε θα ήθελα τώρα να σας δώσω τον λόγο κύριε Υπουργέ και να σας ζητήσω να απευθυνθείτε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. εμφανίζομαι ενώπιόν σας για να σας εξηγήσω τις ε, Βασικέ δραστηριότητε τη Ισπανική Προεδρία σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Οι προτεραιότητε βρίσκονται σε αυτό το έγγραφο και θα σα δοθούν μετά την παρέμβασή μου. Μετά την εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η Ισπανική Προεδρία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο όπω καθορίζεται από τη νέα συνθήκη που επιτρέπει, αφήνει περιθώριο για μεγαλύτερη μεγαλύτερε αρμοδιότητες. Κάτι που δίχω άλλο θα αποβεί υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διευκολύνουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου στις δράσεις που σκοπεύουμε να προωθήσουμε κατά τη διάρκεια των ε, έξι μηνών, πέρα από τις συνήθεις συναντήσεις στην αρχή και στο τέλος της Προεδρίας, δεσμεύομαι να εμφανιστώ και πάλι ενώπιόν σας το Μάρτιο για να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα του Εαρινού Συμβουλίου Μεταφορών. Η Ισπανική κυβέρνηση έχει στόχο να κάνει ένα χρονοδιάγραμμα που θα είναι επικεντρωμένο στην όθηση που θα πρέπει να δοθούν στα προγράμματα και στις δράσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάκαψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, οι στόχοι μας στην, ε, το εξάμεινο αυτό της Ισπανικής Προεδρίας θα επικεντρωθούν στο θέμα της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταφορές θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για να καταστούν περισσότερο βιώσιμε οι οικονομίε μα. Η Ισπανική Προεδρία θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα μέτρα που επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών που καθιστούν πιο αποτελεσματική την κινητικότητα, που βελτιώνουν και επεκτείνουν τα δίκτυα μεταφορά και που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των δικτύων αυτών. Για το λόγο αυτό, με βάση τους προτανατολισμούς όπως διατυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, θα επικεντρωθούμε στις βιώσιμες μεταφορές σε αστικό και μητροπολιτικό πλαίσιο, γιατί εκεί ακριβώς επικεντρώνεται οι περισσότερες αρνητικές πτυχές των μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πέρσι τον Οκτώβριο ένα πρόγραμμα δράσης για την ε, αστική γεννητικότητα. Αυτό αποτελεί μια σειρά από απτές ενέργειες αυτό το πλαίσιο. Η Ισπανική Προεδρία, συνάντηση των Υπουργών που θα γίνει στο Λιακορούνια τον ερχόμενο Φεβρουάριο, θα προσπαθήσει να προωθήσει τα βιώσιμα μοντέλα κινητικότητας στο αστικό πλαίσιο. Ελπίζουμε να μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία έτσι ώστε το Συμβούλιο του Ιουνίου ε, να μπορέσει να υιοθετήσει συγκεκριμένες αποφάσεις. Όπως γνωρίζετε, μετά από την δημοσίευση το προηγούμενο ε, Φεβρουάριο της Πράσινης Βίβλου που αφορούσε την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο ε, Συμβούλιο Μεταφορών της 11ης Ιουνίου υιοθετήθηκαν ορισμένες αποφάσεις που καλούν την Επιτροπή να, εφαρμο, πάρει δύο πρωτοβουλίε. Να υποβάλει μια πρόταση αναθεώρηση του προσανατολισμού του δικτύου πριν από το 2010 και να προετοιμάσει μια ανακοίνωση για τα κριτήρια που θα καθορίσουν τη νέα απόφαση για τι αρχέ του 2010. Η Ισπανική Προεδρία έχει στόχο να συμβάλλει έτσι ώστε τα σχόλια του Συμβουλίου θα θεωρηθούν ως σημεία αναφοράς. Τα βασικά θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα ε, πάνω στην οποία θα στηριχθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Αποφασίσαμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσουμε στη Σαραγκώσα τις επόμενες μέρες, ε, ε, στο μέλλον στις 8 και 9 Μαΐου, μία συνάντηση για να αναλύσουμε το θέμα των διευρωπαϊκών μεταφορών. Μόλις καθορίσουμε τη μεθοδολογία θα περατωθεί η διαδικασία αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού, ε, Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή, η... Η Ισπανική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στον αποκαλούμενο ευρωπαϊκό διάτρομο. Είναι όμως πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την ε, σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων λόγω των θετικών οικολογικών τόσο που έχει. Όπως ξέρετε, ε, υιοθετήθηκε τον Ιούνιο μία απόφαση για ένα νέο κανονισμό που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των, ε, ε των συνδρομικών μεταφορών. Το εξάμεινο λοιπόν της Ισπανικής Προεδρίας θα προσπαθήσουμε να λάβουμε μια συμφωνία, ε, να υπάρξει μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να μας απασχολήσει και η ποιότητα των απαρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία εγγύηση των δικαιωμάτων των επιβατών. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία συμφωνία που θα αφορά τα δικαιώματα των επιβατών για συλλογικές μεταφορές, χερσαίες μεταφορές και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Έχουμε πρόθεση να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Μεταφορών σε μια προσπάθεια να προωθήσουμε αυτούς τους κανονισμούς. Η Ισπανική Προεδρία θα συντονίσει τις, ε, τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να καταλήξει σε μια ικανοποιητική συμφωνία η οποία εγγυάται τα ίδια δικαιώματα σε όλους τους χρήστες μεταφορών μεταφορικών μέσων, συγχωρείτε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δούμε διεξοδικότερα το θέμα της αναγνώρισης του δικαιώματος των επιβατών στην ενημέρωση. Πάρα πολύ συχνά δεχόμαστε διαμαρτυρίες από πολλούς επιβάτες. Είναι επίσης σημαντικό να προχωρήσουμε τις εργασίες μας σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινοτική λύση σε περίπτωση προστασίας των καταναλωτών, ε, για την προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση πτώχειας της μιας αεροπορικής εταιρείας. Αυτοί οι δύο τομείς θα μας απασχολήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εναέριες μεταφορές, έχουμε σκοπό να προωθήσουμε τους ενιαίους ε, ουρανού, ευρωπαϊκούς ουρανούς, ουρανούς που αποτελέσουν με έναν ακρογωνιαίο λίθο γιατί θα επιτρέψει μεγαλύτερη ασφάλιση διάσκεψη της Μαδρίτης που θα, ναι, από την που θα οργανωθεί στις 25-26 Φεβρουαρίου θα πρέπει να αποφασίσει για ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα καταλήξει στη δεύτερη φάση του 2012. Θα πρέπει να υιοθετηθούν τα μέτρα που θα επιτρέψουν την πρακτική εφαρμογή του δεύτερου νομοθετικού πακέτου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε τι τρόπο θα μπορούσαν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Σε ό,τι αφορά την βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα των θαλασσίων μεταφορών, θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εγκριθεί η οδηγία που καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική ε, διαβίβαση των στοιχείων των στοιχείων που θα πρέπει να δίνουν ε, τα ε, ε, σκάφη κατά τον απόπλου και τον κατάπλου σε ένα λιμένα, από ένα λιμένα. Πάρα πολλές φορές οι διατυπώσεις δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Η ενδυνάμωση του τομέα των μεταφορών είναι ένας άλλος από τους στόχους της Προεδρίας μας. Γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο διακήρυξης για το έγνο που επιτρέπει τη συνέχισή του και μετά το 2013. Το πρόγραμμα Γαλιλαίο, τρία σημεία. Θα θέλαμε να γίνει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του προγράμματος. Προβλέπεται η έγκριση της τροπολογίας του κανονισμού, ο οποίος διέπει τον ε, οργανισμό ε, του Γκαλιλαίου και ε, έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε τρία κέντρα ελέγχου που αποσυμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο του Νοέμβριο του 2007 τα συστήματα μεταφορών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα δράση που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2008, έχουμε σκοπό Λοιπόν να καταλήξουμε στο οριστικό κείμενο τη οδηγία για τα φύση συστήματα μεταφορών ε, και αυτό σε ό,τι αφορά τις σχέσε μεταφορές. Ήδη έχει υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ένα άλλο θέμα, μια άλλη προτεραιότητα για τις ε, εργασίες μα αφορά την εγγύηση της ασφάλεια για όλους τους τρόπους ε, μεταφορά. Και πραγματικά η Προεδρία θα είναι απόλυτη σε αυτό το τομέα σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχει μια ε, αναθεώρηση των κανονισμών ε, σε ό,τι αφορά τις έρευνες σε περίπτωση ε, δυστυχήματος. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ανακριτικών αρχών και θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη στήριξη στα θύματα και στους ε, συγγενεί του. θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση της διαβίβασης του καταλόγου των επιβατών στην αρμόδια αρχή. Στα πλαίσια τη ε, οργάνωσης ε, της ε, διεθνούς ε, αεροπορίας θα υποβληθεί πρόταση στο Μοντρεάλ στις 29, 30 και 31 Μαρτίου για να υπάρξει μια παγκόσμια δράση που θα οδηγήσει σε μια βελτίωση, σε βελτίωση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πιλότων και των αρχών ελέγχου. Πάρα πολύ συχνά οι πολίτες ε, ανησυχούν και στην Λακορούνια θα υποβάλω στους συναδέλφους μου το πρόβλημα αυτό που αφορά την ασφάλεια στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η Ισπανική Προεδρία συμφωνεί ότι υπάρχει ανάγκη να λαμβάνονται με διαδικασία δυνατόν να μπορούμε να επιτύχουμε μια συμφωνία για τόσο σημαντικά θέματα. Λόγω τη σημασία που έχει κοινωνικό επίπεδο, οι αποφάσεις σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Οι Ευρωπαίοι πολιτε δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να μπορούμε να επιτύχουμε μια συμφωνία για τόσο σημαντικά θέματα. Λόγω τη ε, σημασια που έχει σε κοινωνικό επίπεδο η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό σημείο στο χρονοδιάγραμμα <clears throat> τη ευρωπαικη πολιτικη Η Ισπανική Προεδρία θα υποβάλει προτάσεις για το θέμα των μεταφορών. Ε, και αυτό και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δράση για την περίοδο 2011-2020. Σε αυτό το πλαίσιο θα οργανώσουμε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου και γενικών διευθυντών μεταφορών στη Μαδρίτη τον ερχόμενο Μάιο και θα ασχοληθούμε με την κουλτούρα της ασφάλειας μέσα στις επιχειρήσεις. Η Ισπανική Προεδρία θα υποβάλει τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Το εξάμεινο αυτό θα θέλαμε να προωθήσουμε και τις σχέσεις μα με τις τρίτες χώρες. Η βασική προτεραιότητα αφορά τη διαπραγμάτευση της δεύτερης φάσης διαπραγματεύσεων ε, για την ε, ασφάλεια των μεταφορών ε, τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 13 Ιανουαρίου πήγα στις Ηνωμένε Πολιτείες για να πάρω σε μια συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών Ρέι Λάγουτ. Ο βασικός μου στόχος ήταν να δοθεί μια νέα πνοή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Στη συνάντηση αυτή ενημέρωσε για την ευρωπαϊκή θέση και τόνισα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια εξισορροπημένη συμφωνία έτσι ώστε να υπάρχει αμοιβαίο άνοιγμα ε, <clears throat> προς την αγορά. Ο Υπουργό Μεταφορών στι Ηνωμένε Πολιτείε μου είπε ρητά ότι ε, η αποτυχία είναι ε, ένα θέμα που δεν τίθεται καν προς ε, συζήτηση. Ελπίζουμε η συνάντηση στην Παδρίτη θα καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη συμβολή που μας δίνει ο πρόεδρος κύριος ε, Σίμψον. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στη Βραζιλία θα γίνει μια διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Έχουμε πρόθεση κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής να υπογράψουμε μια διμερή συμφωνία για το θέμα της ασφάλειας ασφάλειας, ε, συμφωνία μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παρατηρήσατε κυρίες και κύριοι ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, ε, φιλόδοξο αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αφορά το θέμα της ασφάλειας, των μεταφορών. Ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα, όπως μας απασχολεί ιδιαίτερη σχέση μας με αυτή την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσα να βασιστώ στην υποστήριξη στις προτάσεις και στις προτάσεις και στις υποδείξει όλων των συναδέλφων τη Επιτροπής Μεταφορών που θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, συνεισφορά σας και για την ομιλία σας. Ε, πριν δώσω τον λόγο στον συντονιστή, συντονιστές να σας διαβεβαιώσω πως ε, χάρηκα που άκουσα την αποφασιστικότητά σας ε, για να εμπλακείτε στην συμφωνία την αεροπορική Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόθεση του νέου γύρου διαπραγματεύσεων το Φεβρουάριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σας ευχαριστώ που προσωπικά ενδιαφέρεστε για αυτό το ζήτημα. Και ελπίζω κύριε Υπουργέ να είμαι στη Σαραγώσα τον Ιούνιο. Ελπίζω να τα καταφέρω Καθώ Καθώς ε, μου λέει η κυρία Γέλα Σέντερ είναι ωραίο κομμάτι της Ισπανίας. Ε, κύριε Πρόεδρε και εσείς ε, και, και οι άλλοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον συντονιστή του ΕΛΚ, τον κύριο Γκρός. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις δηλώσεις στα δικά μου τα μάτια ήσασταν πολύ πιο συγκεκριμένο από αυτά τα οποία διαβάζαμε και ακούσαμε εδώ πέρα. Δείξατε σημάδια πως θέλετε σε σημαντικούς τομείς να δώσετε κάποια μηνύματα και βεβαίως ε, κάποιοι φάκελοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς εδώ πέρα, θα το πούν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά γνωρίζω πως ε, άλλες προτεραιότητες έχει το Συμβούλιο αλλά ελπίζω να έχουμε έναν ίδιο ρυθμό σε κάποια σημεία για να μην οδηγηθούμε σε ρυθμία. Η αηφορία είναι σημαντική ειδικά στις αστικές ε, συγκοινωνίες ε, σε αυτή την επιτροπή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα καθώς ε, θα φτάσουμε συνολικά 80% του πληθυσμού να κατοικεί σε αστικές ζώνες, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της κινητικότητας, οπότε το ερώτημά μου είναι θεωρείτε πως αυτή η ήπια πολιτική της ανταλλαγής των καλών μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης και τα λοιπά επαρκεί ή θεωρείτε πως πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα εμείς βεβαίω υποφέρουμε στη χρηματοδότηση. Ιδέες υπάρχουν, καλά έργα υπάρχουν, υπάρχει και ένας κατάλογος προτεραιοτήτων. Ποιες είναι όμως οι προτάσεις του Συμβουλίου έτσι ώστε αυτά που λέμε θεωρητικά να μεταφραστούν σε κάτι το πρακτικό. Ποια είναι τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο με την Κομισιόν ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη αντίφαση που λένε πολλά ωραία πράγματα οι Υπουργοί Συγκοινωνιών και μετά έρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών και τελειώνει το παραμύθι εκεί πέρα. Συγκεκριμένες λοιπόν ιδέες ε, ε, για την σύγχρονη τεχνολογία συμφωνούμε μαζί σας 100% βλέπω και εγώ βεβαίω Εντάξει, η οδική κυκλοφορία αναφέρεται κάπως λιγότερο, αλλά ακριβώς σε αυτό τον τομέα νομίζω, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, θα δούμε στο μέλλον ε, καλύτερη ξύλιση και αν προβλεφθούν βέβαια στα απαραίτητα κονδύλια. Έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους καθαρούς κινητήρες και να έχουμε και συγκεκριμένα νούμερα και να προωθήσουμε την έρευνα. Ε, νομίζω αυτό θα αποτελούσε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ευρώπης και για το μέλλον. Νομίζω και αυτό θα καθόριζε και την Ευρώπη παγκοσμίως, δηλαδή έρευνα ναι αλλά με τι μέσα. Και είστε διατεθειμένος να ορίσετε νούμερα στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπάρχουν ε, επίσης ε, και πολλοί στόχοι για διεθνείς συμφωνίες, τους αναφέρατε. Πράγματι, ειδικά στην ε, ναυτιλία είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το αναφέρατε δίπλα στην αεροπορία, πως δεν είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, αλλά πρέπει να κινηθούμε σε διεθνές επίπεδο, αλλιώς θα χάσουμε την αξιοπιστία μας, γιατί βεβαίως θα πάνε χαμένοι και οι κόποι μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπετε σημαντική πρόοδο στον τομέα της ε, ναυτιλίας. Αναφέρατε ήδη κάποια πράγματα για την αεροπορία. Και μια τελευταία ερώτηση που φαντάζομαι θα την θέσουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Για το θέμα εσωτερήκευση του κόστους, η Σουηδική Προεδρία μας είπε πώς γίνεται μία μελέτη για την Ευρωβινιέτα και τις επιδράσεις της ε, και μετά δήλωση που μας είπε ότι δεν θα ασχοληθεί με το θέμα. Γνωρίζετε πως έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Να ρωτήσω γιατί δεν αναφέρατε αυτό το ζήτημα σήμερα. Γνωρίζω πως ε, θέλετε να έχετε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Πώς φιλόδοξοι θα είστε σε αυτό το τομέα. Ε, ευχαριστώ κύριε Γκρός. Να πω πως ε, θα ήθελα οι συντονιστές να μιλήσουν τέσσερα λεπτά, μετά τρία λεπτά οι βουλευτές για να απαντήσει και ο κύριος Υπουργός. Και κύριε Υπουργέ, νομίζω μπορείτε να απαντήσετε σε τρεις-τρεις ερωτήσεις για να μην συσσωρευτούν πάρα πολλέ. Ο κύριος Αλχαντραουή για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω πρώτα απ' όλα, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία δεν έχω αμφιβολία πως ε, εσείς ε, προσωπικά θα εμπλακείτε για να μπορέσετε να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα τους ερχόμενους μήνες και θα σας υποστηρίξουμε υπό την προϋπόθεση ότι θα κινηθείτε προς ε, μια πιο φιλόδοξη και καλύτερη πολιτική μεταφορών πράγματα, φιλόδοξο το πρόγραμμα που παρουσιάσατε. Βεβαίω αυτό είναι δύσκολο γιατί το Συμβούλιο κινείται στο ρυθμό του πιο αργού κράτους μέλους και είναι επιτυχία αν μπορέσετε να επιταχύνετε αυτόν τον ρυθμό και να σημειωθεί πρόοδος. Ξέρετε πως είναι σημαντικά τα θέματα γιατί συζητάμε για το μέλλον των μεταφορών, οι προκλήσεις είναι μεγάλες, πρέπει να κάνουμε στρατηγικές επιλογές για το τι θα κάνουμε τα επόμενα 10-20 χρόνια για να οδηγηθούμε σε αποτελεσματικό, κοινωνικό, ασφαλές και αηφόρο σύστημα μεταφορών. Αλλά Ακούμε πάρα πολύ συχνά καλές δηλώσεις από το Συμβούλιο, μιλάει για υφόρες, μεταφορές και τέτοια ωραία πράγματα και τα ακούσαμε και στην Κοπεχάγη, αλλά όταν φτάνουμε στην ε, νομοθεσία την συγκεκριμένη έχουμε περισσότερους δισταγμούς όπως π.χ. με την Ευρωβινιέτα, το ανέφερε και ο κύριος Γκρός για εσωτερικεύση του κόστους, αλλά είναι ένα από τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Και θέλω να ακούσω τι άποψη έχετε. Ε, χαίρομαι που ακούω ότι θέλετε να ενισχύσετε την κινητικότητα. Ξέρετε πως για εμάς αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Επίσης ε, μιλήσατε για μεταφορά φορτίων μέσω του σιδηροδρόμου. Σημαντικό κομμάτι όταν μιλάμε για αηφόρες ε, μεταφορές και για διαδρόμους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα. Ο κύριος Κόχ θα ανέφερε τη χρηματοδότηση των υποδομών. Πρέπει να προετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή το πώς ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Πράγματι και τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να λυθούν τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν κάποιες δικογνωμίες, αλλά νομίζω πως μπορούμε να το προωθήσουμε για την αεροπορία σημαντικό είναι να γίνει έρευνα για τα ατυχήματα, να, να σημειωθεί εκεί πέρα πρόοδος για την ασφάλεια να υπάρξει επιτέλους μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν μπορεί ορισμένα κράτη-μέλη να πάρουν μόνο μέτρα. Δεν μου φαίνεται σωστή η ιδέα αυτό. Και αν βρείτε κάποιες λύσεις θα σας στηρίξουμε. Τέλος, οδική ασφάλεια πολύ μεγάλη προτεραιότητα για την ομάδα μου. Η Κομισιόν οπωσδήποτε θα έχει ένα σχέδιο δράσης. Ελπίζω το Συμβούλιο να είναι φιλόδοξο γιατί έχουμε γύρω στους 40.000 νεκρούς ε, το, το έτος και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μέσω του συντονισμού κάποια πρόοδο. Αυτά από εμάς. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δεν θα συμφωνούμε πάντα, αλλά Νομίζω πως αν συνεργαστούμε θα είμαστε πιο ε, ισχυροί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αλχαντραούη. Η κυρία Μάρη στην έργεια του Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας ε, και αναμένουμε και καλή συνεργασία μαζί σας. Αναφέρατε διαφορετικά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις μεταφορές. Ένα δεν αναφέρατε, το οποίο είναι σημαντικό για εμάς φιλελεύθερους την εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις συγκοινωνίες. Γνωρίζουμε πως η εσωτερική αγορά είναι η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς μεταφορές δεν λειτουργεί. Γι' αυτό αυτό το οποίο αποφασίστηκε το 1992 επιτέλους να δημιουργηθεί, δηλαδή η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Τι σκοπεύετε, τι, θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει. Σημαντικά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά βεβαίως πρέπει να συμφωνήσουν και οι χώρες να τηρούν τα συμφωνημένα. Να μην οδηγούμαστε σε προστατευτισμό, αλλά αμοιβαία να υπάρχει ε, να μπορεί να βαστεί ο ένας τον άλλον και είτε μιλάμε για το καπατάζ είτε μιλάμε για τις εμπορευματικές μεταφορές στους σιδηροδρόμους. Το επόμενο θέμα είναι η αηφορία το αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε πως υπάρχει και βλάβη του κλίματος από τις συγκοινωνίες και πρέπει να εξελιχθούν οι συγκοινωνίες. Τι βάρος δίνεται στην έρευνα και στην καινοτομία. Είναι σημαντική πτυχή ε, στο τομέα των συγκοινωνιών. Και τρίτον αναφέρεται την ασφάλεια των ε, πτήσεων ως ε, προτεραιότητα. Ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα σκάνερ, τους ανιχνευτές υγρών και τους σαρωτές σώματος, ειδικά μετά το περιστατικό που έγινε και στο Μόναχο. Αναρωτιόμαστε αν αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή ε, επαρκούν στα αεροδρόμια, αν πως χρειαζόμαστε ένα άλλο σύστημα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Και το ερώτημα είναι, οι σαρωτές μπορούν να μας δώσουν αυτή την ασφάλεια, χρειαζόμαστε άλλες δυνατότητες. Δικαιώματα των επιβατών τα αναφέρατε. Υπάρχουν και διάφορες εκθέσεις σχετικές τις οποίες συζητάμε. Ξέρετε πως μιλάμε και για τις συγκοινωνίες με πούλμαν και για τα πλοία. Νομίζω θα έχουμε καλή συνεργασία σε εκθέσεις που εκκρεμούν. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στην ε, εσωτερική του εξωτερικού κόστου που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες και εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μια λύση και ε, έστω και αν δεν είναι η πανάκια ε, όπως λέει ο κύριος Σελχαντραουή πρέπει νομίζω να προχωρήσουμε και θα ήθελα να μάθω την άποψή σας και κάτι άλλο το οποίο αφορά εμένα ιδιαίτερα πάρα πολύ για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Εσείς ειδικά ως Ισπανός που βρέχεστε από παντού από θάλασσα νομίζω πως θα δώσετε βάρος αν και δεν το αναφέρατε ρητός. Ποια είναι η άποψή σας για, την, ε, για τις συγκοινωνίες της ε, θαλάσσιες και την ε, πολιτική που έχουμε ακολουθήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε ή πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Το τελευταίο μου ερώτημα αφορά τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι στην Επιτροπή μας. Τι, α, μακρηγόρησα. Όχι, απλά να δώσουμε και την ευκαιρία στον κύριο Υπουργό να μιλήσει. Λοιπόν, θαλάσσια πολιτική τότε παραμένει η τελευταία μου ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Απλά ο Υπουργός Τουρισμού θα έρθει το απόγευμα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Θα θέλατε να απαντήσετε στις συγκεκριμένες αυτές ερωτήσεις και μετά θα δεχτούμε άλλες τρεις. Αν θέλετε απαντήστε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι βουλευτές, όπως και να έχουν τα πράγματα, εγώ είμαι διατεθειμένος να επιμείνω στα θέματα που απασχολούν περισσότερο την Επιτροπή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα που μου ετέθησαν. Υπάρχει ένα θέμα που ανακύπτει συνέχεια και που αφορά το πρόβλημα των δυστυχημάτων. Σε αυτό αναφέρθηκε ο πρόσωπος της σοσιαλιστικής ομάδας. Η Ισπανική Προεδρία πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το επίπεδο ασφάλειας. Και αυτό αφορά όλα τα μέσα μεταφοράς, αφού ο στόχος μας είναι η Ευρώπη να γίνει από τα ασφαλέστερα μέρη μετακίνησης στον κόσμο. Μπορούν ότι υπάρχει ένα εναρμονισμένο σύστημα. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η Ισπανική Προεδρία θα ασκήσει πιέσει στο Συμβούλιο για να υπάρξει ένας κανονισμός σχετικά με τις έρευνες μετά από ένα δυστύχημα. Εκεί θα πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο η ανεξαρτησία των εθνικών φορέων, το ρόλο του Οργανισμού ε, Αεροπορικής Ασφάλειας, αλλά και η προστασία και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών <clears throat> που δημοσιεύονται κατά τη διάρκεια των τεχνικών ερευνών. Ορισμένοι βουλευτές και ιδιαίτερα πρόσωπος της ομάδας των φιλελευθέρων, έθεσε το θέμα της ασφάλειας. Μετά από όσα συνέβησαν στο Ντιτρόιτ, κάτι που κινητοποίησε όλη τη διεθνή κοινότητα. Μπροστά σε μια τέτοια πραγματικότητα, η δική μας ευθύνη είναι να δώσουμε μια απάντηση που δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας των δικών μας αεροδρομίων. Εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες λύσεις που μας παρέχει η τεχνολογία χωρίς ποτέ να ξεχνάμε την ανάγκη να μειωθούν στο ελάχιστο να μειωθεί στο ελάχιστο η ενόχληση για τους επιβάτες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να επιτύχουμε μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, χωρίς όμως από την άλλη πλευρά να φυγούν τα δικαιώματα των επιβατών. Η Ισπανική Προεδρία θα πρέπει να υιοθετήσει μέτρα που θα πρέπει να βασιστούν σε μια ευρεία συνένεση. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να γίνει αυτό. Η Ισπανική Προεδρία έχει σκοπό να εργαστεί σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια συμφωνία στο Συμβούλιο. Στη Λακορούνια στις 12 Φεβρουαρίου θα εξετάσουμε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Μεταφορών. Έχω τη βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα καταφέρει να δώσει μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Ξέρω ότι θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσει για την ασφάλεια. Η εγγυήση όμω αυτή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια όκληση για του επιβάτε. Θα πρέπει να βάλουμε τέλο στην ε, ενόχληση ε, των ε, ε, επιβατών ενόχληση που δημιουργείται σαν αποτέλεσμα τη χρήση των διαφόρων συστημάτων ελέγχου. Έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι συνεχίζει, του γεγονότος συνεχίζει να υπάρχει η απειλή ε, της μεταφοράς εκρηκτικών υγρών. Νομίζω ότι αν μειωθεί το επίπεδο των ελέγχων θα μειωθεί και το επίπεδο της ασφάλειας. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμείς είμαστε υπέρ της παράτασης του περιορισμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υγρών στις χειραποσχευές. Δεν έχουμε ακόμα μία τεχνολογία η οποία μας επιτρέπει να δώσουμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. προβλέπεται η υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση των εκπομπών. Η μείωση των εκπομπών είναι ένα θέμα που δεν θα πρέπει μόνο να συζητάμε, αλλά θα πρέπει να μας οδηγήσει και στη λήψη αποφάσεων. Αυτό θα θέλαμε να το τονίσουμε στη συνάντηση που θα γίνει στη Μαδρίτη και που θα πρέπει να καθορίσει την πορεία που θα ακολουθήσουμε μέχρι το 2012. Η συνάντηση αυτή θα οργανωθεί, όπως είπαμε, στη Μαδρίτη, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί θα υπογραμμίσουμε το θέμα της πληροφόρησης. Διατυπώθηκαν μερικές ερωτήσεις για θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Καταρχάς, ο πρόσωπος της ομάδας ε, του ΕΛΚ, αλλά και άλλοι βουλευτές, διατύπωσαν ερωτήσεις σχετικά με την αποκαλούμενη ευρωβινέτα και το εξωτερικό κόστος των μεταφορών. Έχω απόλυτη συνείδηση της σημασίας που έχει αυτό το σημείο, καθώς και θέματα που αφορούν τη συμφόρηση, το θόρυβο κτλ. Θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι η προηγούμενη Προεδρία κατάφερε να καταλήξει σε κάποια συνένεση σχετικά με τα τόσο ευαίσθητα αυτά προβλήματα. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προσκόμματα στην αρχή της εφαρμογής ο, Ριπένον ο πληρώνει. Το αντίθετο. Θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα του υπολογισμού του κόστους. Αυτό θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τη διπλή φορολογία ή τον αθέμητο ανταγωνισμό. Η παρούσα χρήση θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία ακριβώς για αυτό το λόγο γιατί θα μπορούσε να υπάρξει μια μείωση τη ανταγωνιστικότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε στη διάθεσή μα συγκεκριμένε αξιολογήσει που αφορούν το κόστο που θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή μια νέα οδηγία. Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία, έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε να συζητάμε την πρόταση οδηγία σε τεχνικό επίπεδο και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τι διάφορε συγκρούσει. Θα πρέπει όμω να λάβουμε υπόψη μα το κόστο που συνεπάγεται η διάκριση μεταξύ ιδιωτικών, ε, αυτοκινήτων ιδιωτικής και εμπορικής χρήσης. Θα οργανώσουμε και μια τεχνική συνάντηση για το θέμα αυτό με τον ε, ε, τεχνική συνάντηση. Ο Επίτροπος Κάλλας είπε ήδη ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τον από πλευρά της Βελγικής Προεδρίας όταν πλέον θα έχουν επιληθεί τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε θα προσπαθήσω να απαντήσω και στα άλλα ερωτήματα. Θα πρέπει να πω ότι η ασφάλεια των αεροπορικών και των σερκιστέρων μεταφορών είναι μια απόλυτη προτεραιότητα. Θα πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει σε ό,τι αφορά τα δυστυχήματα θα οργανώσουμε μια συνάντηση γενικών διευθυντών στη Μαδρίτη για να μπορέσουμε να εξετάσουμε εκτενέστερα αυτό το θέμα και έχω τη βεβαιότητα ότι σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα υπάρχει ευρύτατη συνένεση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταφοράς προϊόντων, αγαθών, θα πρέπει να πω ότι η μεταφορά εμπορευμάτων είναι έμονη ιδέα για μένα η δημιουργία ανταγωνιστικής μεταφοράς εμπορευμάτων και βιώσιμης μεταφοράς. Η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί επαρκώς αφού, αν δεν υπάρχει μια υποδομή η οποία παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ξεπεραστούν δυσκολίες όπως ε, ε για ε, παράδειγμα μία ανεπαρκής σύνδεση μεταξύ των σιδηροδρομικών υποδομών και των άλλων μέσων μεταφοράς. Η Ισπανική Προεδρία δίνει προτεραιότητα στην πρόταση κανονισμού για ένα ανταγωνιστικό σιδηροδρομικό ευρωπαϊκό δίκτυο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ελπίζει σε δεύτερη ανάγνωση με το Κοινοβούλιο να επιτευχθεί μια συμφωνία. Δύο τελευταίες απαντήσεις κύριε Πρόεδρε. Και θα τελειώσω. Μην αρχίσετε να με απειλείτε με το σφυράκι σας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε περαιτέρω, ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε όθηση στις θαλάσσιες μεταφορές για την Ισπανική Προεδρία. Θα δεχτεί με χαρά προτάσεις που έχουν σχέση με τη συνολική βιωσιμότητα των, ε, των μεταφορικών μέσων. Ο πρόσωπος του ΕΛ και της Σοσιαλιστικής Ομάδας μου έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των μεταφορών μας. Θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με το στόχο που εξέφρασε ο Επιτροπός Κάλλας, δηλαδή την ανάγκη από τη μία πλευρά να διατηρηθούν οι επενδύσεις, γιατί οι παραγωγικές επενδύσεις δημιουργούν απασχόληση και οικονομική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι είναι αναγκαίο από αυτή την άποψη, να υπάρξει η δημιουργία ενός ταμείου για τις μεταφορές αυτό είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο. Είμαι σύμφωνο, μίλησε γι' αυτό και ο Επίτροπος Κάλλα και δίχως άλλο έχει τη δική μου στήριξη. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Οπωσδήποτε οι συνάδελφοι θα σα υποδεχθούν σωστά. Λοιπόν, Έχουμε πολλούς συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν και οι δύο συντονιστές θα έχουν τον ίδιο χρόνο με τους υπόλοιπους. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ πρώτα απ' όλα για τους πράσινους και μετά ο κύριος Ζέιλε. Ε, ο κύριος Κράμερ για τους πράσινους. Ευχαριστώ και για αυτά τα οποία μας είπατε. Τονίσατε την αηφορία, αλλά βεβαίω κανένα πολιτικό κόμμα πλέον δεν την παραλείπει. Οπότε συγκεκριμένα έχει από το 1990 αύξηση κατά 30% των εκπομπών η κυκλοφορία. Έχουμε δώσει δισεκατομμύρια για να επιτύχουμε μια μερική μείωση στις κατοικίες και τη βιομηχανία. Θέλετε να ορίσετε ένα στόχο για τις συγκοινωνίες μέχρι το 2020. 20% πρότεινε το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, 10% 30%. Ποιος είναι ο στόχος σας, θέλετε κάποια μείωση για, την, ε, για τις συγκοινωνίες. Στην αστική συγκοινωνία. Όλοι θέλουμε να την προωθήσουμε, αλλά έχουμε την επικουρικότητα. Η μοναδική δυνατότητα να επέμβουμε είναι από τον προϋπολογισμό. Αποφασίσαμε στο Κοινοβούλιο πως τουλάχιστον 40% των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα πάνε στο σιδηρόδρομο, ενώ για τις συγκοινωνίες. Μέχρι στιγμής πάνε 60% στις ε, δρόμους. Το μπλοκάρει το Συμβούλιο θα δεσμευτείτε πως τουλάχιστον 40% των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα πάνε στο σιδηρόδρομο για να αναγκαστούν και οι πόλεις ε, και τα κράτη βεβαίως να μην χτίζουν μόνο δρόμους. Κατόπιν, Ευρωβινιέτα. δεν θα υπάρξει αδικία εάν την εγκρίνουμε. Υπάρχει τώρα αδικία στον ανταγωνισμό. Ξέρετε πως στο σιδηρόδρομο κάθε ε, αμαξοστοιχεία πρέπει να πληρώσει διόδια. Στον αυτοκινητόδρομο όχι. Έχουμε την κατάσταση στην Ισπανία πως ε, ήταν συνέχεια ε, δεν βλέπαμε καθόλου φορτηγά στους ισπανικούς αυτοκινητόδρομους και πηγαίναν όλοι και είχαν μπλοκάρει τους επαρχιακούς δρόμους γιατί δεν πλήρωναν εκεί διόδια. Τι θα γίνει με αυτό. Επίσης θέλετε να προωθήσετε την μεταφορά αγαθών με, με το σιδηρόδρομο. Είστε υπέρ της κυκλοφορίας των Gigaliner και στην υπόλοιπη Ευρώπη πριν Σκανδιναβίας. Γιατί εκεί πέρα θα σκοτώσουμε το σιδηρόδρομο. Θα πάνε όλα στα φορτηγά. Ποια είναι η θέση σας. Γιατί απειλείται και η μεταφορά σε αγαθών από το σιδηρόδρομο και στην Ισπανία. Επίση δικαιώματα επιβατών και εκεί πέρα υπάρχει αδικία. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε. Στο σιδηρόδρομο ε, έχουμε μετά από δύο ώρες 50% ε, αποζημίωση. Στη ιδέα αεροπορία πρέπει να περάσουν πέντε ώρες για να δοθεί αποζημίωση. Θέλετε να το προωθήσετε ίδια δικαιώματα για όλους. Τέλος, οδική ασφάλεια. Και εδώ πέρα μπορείτε να τονίσετε την αηφορία. Στις 26 χώρες έχουμε όριο στον αυτοκινητόδρομο πλην μίας. Θέλετε να υπάρξει όριο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να προωθεί η ασφάλεια και οι εκπομπές. Ε, λοιπόν που το λέω, η χώρα αυτή βεβαίω που δεν έχει όριο στον αυτοκινητόδρομο είναι η Γερμανία, η δική μου. Κύριε Ζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την δέσμευση που επιδεικνύεται. Εγώ έλαβα απαντήσεις σε ερωτήσεις μου ήδη. Οπότε θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι είστε υπέρ της ασφάλειας στην αεροπορία και για το ότι σκοπεύετε να συνάψετε συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Βεβαίως θα μιλάμε για τις υδροδρομικές μεταφορές. Δεν θα είμαι εγώ τόσο εκφραστικός όσο ο κύριος Κράμερ, ο συνάδελφος, αλλά βεβαίως πρέπει να σε ευχηθώ επιτυχία όσον αφορά στην αύξηση της διαλειτουργικότητας, και της ε, ασφάλειας και μιλώντας τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και ελπίζω πως θα μπορέσετε και εσείς να βελτιώσετε κάπως την κατάσταση. Τώρα μιλώντας για τα δικαιώματα όμως των επιβατών συγκεκριμένα για τα πλοία και ε, τα λεωφορεία Υπάρχει κάτι το πολύ πρακτικό πέρα από την νομοθεσία. Ένα πράγμα ενδιαφέρει τους ανθρώπους. Τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε τα εισιτήρια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σιδηροδρομικά εννοώ, να πολλούνται οπουδήποτε. Να είναι ένα δηλαδή το εισιτήριο ενιαίο. Και ε, κάναμε μια έρευνα πως δεν θα υποφέρει και ο κλάδος ε, εάν μειωθεί ε, το επίπεδο θορύβου που ε, κάνουν οι μεταφορές. Και εάν δεν κάνουμε τίποτα για την Ευρωβινιέτα, εντάξει, εξακολουθεί να, να υπόκειται στην επικορικότητα ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους βουλευτές να με βοηθήσουν να τελειώσουμε 12.30. Κύριος Δεκάνατης Φασκουάλ. Και δύο, δύο λεπτάκια ο καθένας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που σκοπεύετε να βασιστείτε μαζί σας. Θα αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις στην Προεδρία σας γιατί έχουμε μια νέα συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας που ισχύει και θα πρέπει να εγκρίνετε μια σειρά από νέα προγράμματα επίσης. Αναφέρθηκε η οδηγία για την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών για τους επιβάτες. Μας είπατε ότι επιθυμείτε ένα συνενετικό αποτέλεσμα. Όντως, είναι σημαντικό να εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση και με σημαντική συνένεση. Επίσης, κατανοώ ότι πρέπει να έχετε ρεαλιστικούς στόχους για την, το εξάμεινο της Προεδρίας σας. Ενδιάμεση αναθεώρηση, διευρωπαϊκά δίκτυα. Σας στηρίζουμε απολύτως σε αυτά, όπως επίσης και για τον, τη Μεσογειακή Οδό. Το πολύ σημαντικό θέμα όμως είναι η αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων και θα χαρούμε πολύ αν μπορέσετε να ασχοληθείτε και να ολοκληρώσετε το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Επίσης, φιλόδοξη στόχη και για την ασφάλεια στα αεροδρόμια. Και εκεί πρέπει να ληφθούν συνενετικά οι αποφάσεις. Έχουν γίνει διάφορες δοκιμές πιλωτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ε, ΙΠΑ, αλλά τα αποτελέσματα είναι λίγο περίεργα. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις και να τις βρούμε συνανέτικα. Όσον αφορά τώρα τους υδροδρόμους, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ναι, πρέπει να έχουμε καλές οδικές μεταφορές, χρειάζονται για την εσωτερική αγορά, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται πέρα από αυτό. Επίσης, Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που ενθαρρύνετε τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα γιατί είναι περιορισμένα τα δικά μας κονδύλια και μπορούν να μας ενισχύσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, κύριε κυρία Αλβάρες, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό. Χαίρομαι που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα ασφαλείας. Γνωρίζω ότι το Υπουργείο σας αλλά και η Προεδρία παίρνει πολύ σοβαρά το θέμα αυτό. Μου άρεσε ιδιαίτερα η πρότασή σας για μεταρρύθμιση του συστήματος έρευνας ατυχημάτων, κάτι που θα μπορούσε και να βελτιώσει τις έρευνες, αλλά παράλληλα να σέβεται την ιδιωτικότητα των οικογενειών. Όσον αφορά τώρα τα συστήματα ασφαλείας στα αεροδρόμια αυτά τα συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν καθυστερήσεις, μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση κάποιους επιβάτες, οπότε περιμένουμε να ακούσουμε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορέσετε να προστατεύσετε τα δικαιώματα των επιβατών. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε σε πέντε λεπτά τις τέσσερις ερωτήσεις ε, που ακούστηκαν. Δυστυχώς πρέπει να ζητήσω και από εσάς κάποια πειθαρχία. Ευχαριστώ. Δύο βουλευτές ε, διατύπωσαν την ίδια ερώτηση και η ερώτηση αυτή αφορά την ενημέρωση των επιβατών. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των επιβατών, Πιστεύω ότι με την έγκριση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις υδροδρομικές και εναέριες μεταφορές και με την έγκριση της ε, οδηγίας για τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις μαζικών μεταφορών θα έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να πάμε ακόμα πιο πέρα. Οι αερομεταφράσει ήταν οι πρώτε που αποτέλεσαν αντικείμενο αυτού του κοινοτικού κανονισμού. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε τα συστήματα πληροφόρηση. Καταρχά, υπάρχει υποχρέωση να ενημερώνονται διαρκώ οι επιβάτε για την κατάσταση και για τα προβλεπόμενα ωράρια αναχωρήσεων, όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν μεταξύ των άλλων και την ε, ακύρωση πτήσεων. Θα πρέπει να επιμένουμε στις ε, αεροπορικές εταιρείες και να τονίζουμε ότι θα πρέπει να ε, ενημερώνουν διαρκώς τους επιβάτες για να μειωθεί η ζημία που θα υποστούν σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης μιας πτήσης. Σε ό,τι αφορά άλλα θέματα Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τεγκράν. Εγώ είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός ταμείου για τις υποδομές. Συμφωνώ και για τον καθορισμό κριτηρίων για μια δημόσια ιδιωτική συγχρηματοδότηση με στόχο τη δημιουργία κινήτρων για τον τομέα των υποδομών. Θα έπρεπε βεβαίως να κινητοποιηθούν πολύ περισσότεροι πόροι. Και ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομία μας διανύει μια δύσκολη περίοδο. Σε ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, συμφωνώ μαζί σας και αναλαμβάνω τη δέσμευση ότι στη συνάντηση της Σαραγκώσα θα υπάρξει μια δήλωση στην οποία με απόλυτα ακριβή τρόπο θα ορίζεται η μεθοδολογία και τα κριτήρια αναθεώρησης. Κατά την άποψή μου αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα που απαιτεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Κατά την άποψή μου θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε με ηρεμία, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς μπροστά σε τέτοιες απειλές. Υπάρχουν Υπάρχει το δικαίωμα της ασφάλειας και υπάρχει το δικαίωμα υποχρέωση προστασίας των επιβατών. Και θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στον τομέα της ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε και τις σημείες που πολύ συχνά προκύπτουν στα αεροδρόμια. Να εγγυηθούμε την ασφάλεια και να εγγυηθούμε ότι δεν θα προκύψει κάποια ενόχληση για τους επιβάτες. Ελπίζω στο, συνέδριο της, ε, στο Συμβούλιο της Λακορούνια θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Θα πρέπει να υπάρξει συνένεση, γιατί δεν έχει νόημα κάθε χώρα να ορίζει τα δικά της κριτήρια ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του συναδέλφου από τους πράσινους, θα ήθελα να τονίσω ότι οι αηφόρες μεταφορές είναι οι μοντέρνες μεταφορές και προς τα εκεί στοχεύουμε. Συνεπώς είμαι υπέρ του να καταβάλουμε προσπάθεια για να αλλάξουμε τον προσανατολισμό των κονδυλίων, δηλαδή να δοθεί προτεραιότητα στις μεταφορές, στις ηροδομικές μεταφορές. Να σας αναφέρω ένα συμβάν στο Υπουργείο μου φέτος το 50% των προπολογισμού αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Αυτό σαν αποτέλεσμα των επιλογών του προκατόχου μου στο Υπουργείο. Σαφώς λοιπόν είναι υπέρ μια τέτοια επιλογής γιατί πιστεύω ότι όλο και περισσότερο θα πρέπει να μας απασχολεί το θέμα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και πιστεύω ότι η διάσκεψη κορυφής με τις Ηνωμένε Πολιτείες και η συνεργασία μαζί τους θα μας επιτρέψει να ε, μολύνουμε όλο, να ρηπαίνουμε όλο και λιγότερο. Ε, βάζοντας στόχο την αποτελεσματικότητα και την εφορία. Συμφωνώ με τον στόχο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Θα ήθελα να θυμίσω ότι οι μεταφορές είναι ένας από τους τομείς που ρηπαίνουν περισσότερο. Αυτό είναι πάντοτε κάτι που θα πρέπει να έχουμε κατά νου και να καταβάλουμε προσπάθειες συνεπώς για να μειώσουμε, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό των, ε, της ε, εκπομπής ε, των εκπομπών. Ένα άλλο ερώτημα αφορά τα φορτηγά των 60 τόνων. Η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι για να μπορέσει να επηρεάσει τα πράγματα ε, αυτή η στον τομέα της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μία συνένεση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει τροπολογία της οδηγίας που αφορά την κυκλοφορία αυτών των οχημάτων. Από τις μελέτες που έγιναν καταλήγουμε ότι σε επίπεδο ασφάλειας η χρήση αυτών των ε, οχημάτων θα πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς, περιορισμούς ταχύτητας, περιορισμούς ε, χειρισμών, απόστασης ε, μεταξύ των οχημάτων, προαπαιτήσεων για τους, για τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Η κυρία Βιλμπάου. Λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις απαντήσεις σας. Καλή επιτυχία στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Ορισμένες πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Γιατί εδώ στην Ευρώπη σκεφτόμαστε πολύ, αλλά δεν ε, κοιτάμε τόσο την εφαρμογή. Για παράδειγμα, διευρωπαϊκά δίκτυα. Στην προτεραιότητα 3. Το πρόγραμμα 3. Τι πρόκειται να κάνετε προκειμένου να απεμπλακεί αυτό. Το πρόγραμμα 3 για τη σύνδεση Γαλλίας και χώρας των Βάσκων. Και επίσης πώς θα συνδυαστεί αυτό με τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας. Τι θα πρέπει να κάνουμε στα λιμάνια μας προκειμένου να είναι αποτελεσματική αυτή η αυτοκινητόδρομη της θάλασσας. Ναι, μεν συμφωνώ μαζί σας για τα όσα είπατε για την αηφορία, αλλά νομίζω ότι το θέμα αυτό της οδού μεταξύ Γαλλίας και χώρας των Βάσκων είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει σαφής κατάλογος των πιθανών προγραμμάτων στα αυτό όσον αφορά τους σιδηροδρόμους και όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή Υπάρχει σε εξέλιξη οδηγία που αφορά το θέμα του χρόνου εργασίας των οδηγών. Μπορείτε να σχολιάσετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Όλο και αυξάνει ο αριθμός των συναδέλφων που θέλουν να λάβουν το λόγο και όλο και μειώνεται ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας για τις απαντήσεις του Υπουργού. Παρακαλώ όμως, αν κάτι έχει ήδη ερωτηθεί, μην το επαναλάβατε. Σας παρακαλώ. Η ε, κυρία Λίχτεμπεργκερ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εμένα προκύπτουν κάποια ερωτήματα από αυτά τα οποία ακούστηκαν ήδη. Πρώτον, εάν εξακολουθείτε να θεωρείτε πως πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαρωτές σώματες ακόμα και αν υπάρχουν μεγάλες ε, αμφιβολίες για το εάν επιτυγχάνουν πράγματι το στόχο τους κάτι το οποίο νομίζω έχει ξεκαθαρίσει δηλαδή δεν είναι τόσο τεχνικά όριμη εξακολουθείτε να είστε υπέρ είπατε πως είναι κάποια δυσάρεστα πράγματα είναι θέμα αναλογικότητας επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα για ένα κέρδος το οποίο δεν έχει ακόμα αποδειχτεί. Εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση και εμπαρόδο αν ενδιαφέρονταν για τέτοιους σαρωτές το Συμβούλιο έχουμε κάποια παλιά μοντέλα που μας έχουν μείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το πουλήσουμε. Δεύτερον, ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα, για κάθε προεδρία, δυστυχώς εδώ με κρέμασαν οι Σουηδοί τι γίνεται με την Σύμβαση των Άλπαιων. Επιτέλους πρέπει να οριστικοποιηθεί. Οι Ιταλοί φέρνουν αντίσταση. Δηλαδή μεταξύ έτσι μεσογειακών χωρών δεν μπορείτε να τα βρείτε και να ολοκληρώσετε αυτό το έργο γιατί νομίζω πως υπάρχει μια ανάλογη σύμβαση ε, που θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και για τα Πυρηναία. Και τρίτον, όταν μιλήσατε για τον κανονισμό περί υγρών στις πτήσεις που θέλετε να τον διατηρήσετε. Τα υγρά που έχουν μαζί τους οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Μιλάω για τα υγρά, το ενόπνευμα στο αίμα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Μιλήσατε για την εσωτερική ναυσιπλοεία, μιλήσατε για την αηφορία και θέλω εγώ να σας πω πως τη Δευτέρα μιλήσαμε εμείς εδώ για την εσωτερική ναυσιπλοεία και διαπιστώσαμε πως είναι γύρω στο 5% στην Ευρώπη, στη χώρα μου εντωμεταξύ είναι γύρω στο 40% αλλά η ρήπανση είναι πολύ περιορισμένη και οι εκπομπέ είναι γύρω στο 1%. Οπότε είναι ένα πολύ αηφόρο τομέα, φιλικός προς το περιβάλλον. Ταυτόχρονα διαπιστώσαμε σχεδόν ομόφωνα και απευθυνθήκαν προ την Κομισιό να λάβει μέτρα. Γιατί ο κλάδος αυτός έχει προβλήματα, αντιμετωπίζει κρίση αυτή τη στιγμή, έχουν καταρρεύσει οι τιμές ε, και η προσφορά φορτίου. Οπότε στηρίζεται την πλειοψηφία αυτής τη Επιτροπής στην έκκλησή της έναντι της ε, Κομισιόν για να βοηθήσουμε την εσωτερική ναυσιπλοεία και συγκεκριμένα τι θα κάνετε. Δεύτερον, μιλήσατε για ασφάλεια. Αυτό το συνδέουμε και με την ασφάλεια στι οδικές μεταφορές. Στι οδικές μεταφορές έχουμε πάρα πολλές απαγορεύσεις για οδήγηση Σαββατοκύριακο και αργίες ε, διατάξεις και διατάξεις και διατάξεις και είναι δύσκολο να προγραμματίσει κανείς αποτελεσματικά τι γίνεται και δυσκολεύουμε για τη δουλειά των, των οδηγών και δεν προωθούν τελικά την ασφάλεια. Συγκεκριμένο ερώτημα. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι για την εναρμόνιση στην οποία οδηγούμαστε για την απαγόρευση οδήγησης ε, στην Ευρώπη και για να μπορέσουμε να ξαναπάμε σε ένα σύστημα ε, στο οποίο θα έχουμε κάποιες απαγορεύσεις μία-δύο μέρες ε, και ξέρω εγώ την Κυριακή. Σας ευχαριστώ που μείνατε εντό χρόνου. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε και να πάμε στις επόμενες ή να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε. Μετά τον κύριο Βαντάλνο, κύριο Κάντσιαν. Eh, Κύριε Υπουργέ, Ήρθατε σε μια καθοριστική στιγμή για έξι μήνες μόνο, αλλά παρόλα αυτά έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη τον επαναπρογραμματισμό κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό από τη στιγμή που μιλάμε για θέματα μεταφορών. Προηγουμένω αναφερθήκατε σε διάφορες υπηρου, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της Νάπολης και θα σα έλεγα να κοιτάξετε τα πρακτικά. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, Αφρική και πραγματικά θα σας έλεγα να το λάβετε αυτό η υπόψη σας. Στην Επιτροπή αυτή μας απασχολεί το θέμα των βιώσιμων μεταφορών και καταλαβαίνω ότι είστε διατεθειμένος να το εξετάσετε αυτό το θέμα και να κάνετε μία προσπάθεια να προωθήσετε μερικές μεγάλες πρωτοβουλίες. Το θέμα μας είναι ενώπιον της κρίσης τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να τεθεί σε κίνηση η οικονομία. Επειδή είμαι εισηγητής για το θέμα της, των δικαιωμάτων των επιβατών είδα την τελευταία έκθεση του Συμβουλίου η οποία ε, είχε τα απολύτως αναγκαία. Θα ήθελα να μου πείτε ε, μία, ε, θα ήθελα να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένο και με τους χρόνους που έχουν τηρηθεί και με το περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που δεν θα μιλήσουν τελικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Η κυρία Τικάου κατόπιν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Ισπανική Προεδρία γιατί στο πρόγραμμα του τρίου της ε, Ισπανικής, Βελγικής και Ουγγρικής Προεδρίας έχουν σαφές πρόγραμμα για τη στρατηγική του Δούναβη καθώς ξεκινάει αρχές ε, Φεβρουαρίου η σχετική διαβούλευση με μια διάσκεψη θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών εάν σκοπεύετε στις, στα άτυπα συμβούλια να θίξετε το ζήτημα μιας πιθανής επαναξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων για να έχουμε περισσότερα κονδύλια για έργα μεταφορών και αν σε αυτά τα άτυπα συμβούλια έχετε προγραμματίσει συνομιλίες για τη διοικητική συνεργασία, για τη διασύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων για τις οδικές μεταφορές. Και τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω στην σημασία των μεταφορών στην ε, επόμενη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 και εδώ πέρα αναφέρομαι στις δουλειές, στις κοινωνικές συνθήκες για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ κύριο Στέρξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα για την οδική ασφάλεια. Στη Λευκή Βίβλο του 2001 είδαμε πως θέλουμε μείωση των νεκρών κατά 50%. Δεν το έχουμε φτάσει αυτό. Ο συνάδελφός μας ο κύριος Γκρός ε, έχει προετοιμάσει μια έκθεση για τη νέα Λευκή Βίβλο που θέλει το 50% να πάει στο 2015 για να το επιτύχουμε σκοπεύετε να πιέσετε την Κομισιόν να κρατήσει το ποσοστό αλλά και το 2020 να πάμε σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Να. Έχουμε επίσης συγκεκριμένο ποσοστό για παιδιά και βαριά τραυματισμένους. Να μιλάμε δηλαδή μόνο για νεκρούς, αλλά και για όσους μένουν ανάπηρους. Είστε ε, διατεθειμένος να θέσετε αυτά τα ποσά, δηλαδή 40% λιγότερους νεκρούς, 40% λιγότερους βαριά τραυματισμένους και 60% λιγότερα νεκρά παιδιά. Ευχαριστώ. you, Ευχαριστώ. Κύριε Στρεμόσο, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου στο Υπουργό. Χαίρομαι που βρίσκεστε σήμερα μαζί μου. Πολύ σύντομα. Σήμερα η Ισπανία είναι ένα νησί από πλευράς σιδηροδρόμων. Η Ρωσία και η Ισπανία χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα στις ράγες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πείτε μου ότι η προτεραιότητά σας θα είναι να συνδέσετε την ισπανική αγορά σιδηροδρόμων με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά. Κάτι που θα βοηθήσει τις μεταφορές κυρίως φορτίων αλλά και επιβατών. Θα στηρίξετε την ιδέα ενός ευρωπαϊκού διαδρόμου που θα περνάει μέχρι και την, από την Νότια Ισπανία και θα μπορεί να συνεχίζει προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάλα Σαντέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω στους κόλπους μας τον Υπουργό και να κάνω ένα σχόλιο μετά από αυτό που είπε και ο κύριος Τρεμέσο. σε σχέση με τις δεσμεύσεις της Ισπανικής Προεδρίας για τη μεταρρύθμιση των διευρωπαϊκών δικτύων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία καλή αγορά η οποία θα περιλαμβάνει και τα Πυρηναία. Είπατε ότι δεσμεύεστε για τον Μεσογειακό Διάδρομο Μιλήσατε για τη σημασία των μεσογειακών συνόρων. Μιλήσατε και για τις συνδέσεις μέσω της χώρας των Βάσκων. Σας ενδιαφέρει λοιπόν το θέμα, αλλά παραμένει το πανάρχιο τείχος μεταξύ Ισπανίας και υπόλοιπης Ευρώπης που είναι τα Πυρηναία. Πρέπει να υπάρξουν διάδρομοι οι οποίοι μεταξύ άλλων θα είναι πολύ σημαντικοί και για τη σύνδεση της Βόρειας Αφρικής με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές τώρα, είναι σημαντικό οι οδικές μεταφορές να χρησιμοποιούνται έξυπνα. Ελπίζω ότι αυτό θα το τονίσετε στο Συμβούλιο. έτσι ώστε να επιτύχουμε αηφόρες οδικές μεταφορές για το μέλλον. Και σίγουρα είναι σημαντικό να υπάρχει διασύνδεση οδικών μεταφορών με τις σιδηροδρομικές και τις θαλάσσιες εσωτερικές πλωτές μεταφορές. προκειμένου τελικά να αποκτήσουμε ένα πιο αηφόρο σύστημα μεταφορών. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να επαναλάβω ορισμένε απαντήσεις Ενδεχομένως κάποιος ε, βουλευτής ε, ήταν απόν όταν έδωσα ορισμένες απαντήσεις και ενδεχομένως θα πρέπει να απαντήσω και πάλι. Νομίζω ότι ήμουν σαφής ό,τι αφορά τους ε, σαρωτές. Επαναλαμβάνω, εάν κάποια θέση δεν είναι κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωση, δεν μπορεί να είναι χρήσιμη. Δεν θα θέλαμε να συνεχιστεί αυτή η διαμαρτυρία των πολιτών για το θέμα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια και να δημιουργήσουμε πρόσκομα στις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και τα δικαιώματα των επιβατών και οι νέες τεχνολογίες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μία γενική απειλή και γενική θα πρέπει να είναι η απάντηση. Η απάντηση θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το Κοινοβούλιο, από αυτή την Επιτροπή και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε μέσω της πρότασης ε, να βρεθεί μία λύση στην συνάντηση στη Λακορούνια. Αυτή είναι η άποψή μας και είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το τονίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε οτιδήποτε στον οποιονδήποτε. Το θέμα αυτό το συζήτησα και με τους Αμερικανούς. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπίσουμε. Δεύτερον, θα ήθελα να πω και να είμαι απόλυτα σαφής ότι ήδη ανέφερα ότι θα είμαι υπέρ μιας παράτασης σε ό,τι αφορά την απόφαση για τα υγρά, για τη μεταφορά υγρών που υιοθετήθηκε το 2006. Σε ό,τι αφορά τα υγρά και τις επικίνδυνες ουσίες για τις σχεσές μεταφορές, για τις οδικές μεταφορές, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να λάβω υπόψη μου την υπόδειξή σας και όλα αυτά τα θέματα για όλα αυτά τα θέματα θα ενημερώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών στα Πούλμαν, όπως είπα στην παρέμβασή μου, η ανταγωνιστικότητα των τρόπων μεταφοράς εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από την εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών. Η Προεδρία θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι που είπα στην παρέμβασή μου. Εμείς συμφωνούμε με την ιδέα ο κανονισμός αυτός να συζητηθεί παράλληλα με αυτόν τον κανονισμό που αφορά αφορά τους επιβάτες θαλασσίων μεταφορών. Έγινε αναφορά και στη συνθήκη των Άλπων. Συμφωνούμε απόλυτα με τους στόχους αυτής της συνθήκης. Ε, μεταξύ των στόχων είναι και η προστασία του περιβάλλοντος. Ε, αυτό είναι ένα τομέας συνεργασία μεταξύ ορεινών περιοχών. Παρ' όλα αυτά, η στόχη τη σύμβαση αυτή είναι μια πραγματική πρόκληση και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκεράσουμε τα διάφορα οικονομικά και οικολογικά συμφέροντα των διαφόρων χρόνων. Για το λόγο αυτό, η Ισπανική Προεδρία είναι έτοιμη να προωθήσει μια πρωτοβουλία η οποία θα επιτρέψει την επίτευξη προόδου σε αυτό το τομέα. Ωράριο εργασία των αυτόνομων οδηγών. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω των κοινωνικών του διαστάσεων. Στι 30 Μαρτίου το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε ένα γενικό προσανατολισμό σχετικά με αυτό το κείμενο. Έχουμε απόλυτη συνείδηση των δυσκολιών αλλά έχουμε τη βεβαιότητα ότι το Κοινοβούλιο θα προβεί σε μια πρώτη ανάγνωση των γενικών προσανατολισμών όπως έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο του Μαρτίου. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε στην Προεδρία μας να προωθήσουμε αυτή την πρόταση. Με στόχο να υπάρξουν εγγυήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, δίχως παράλληλα να θυγεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ε, μεταφορών τόνισα το πόσο με απασχολούν οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας. Έχουμε απόλυτη συνείδηση του γεγονότος ε, του ότι μπορούμε να εργαστούμε περισσότερο. Δίχως άλλο θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ετέθηκε πάλι το θέμα της ασφάλειας των οδικών μεταφορών. Στόχος είναι να υπάρξει μία μείωση κατά 50% την περίοδο 2001-2010. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε θέματα εθνικά. Υπάρχουν χώρες που σεβάστηκαν ε, αυτό το στόχο. Η Ισπανία μείωσε κατά 10% τον αριθμό των θυμάτων ε, τροχαίων σε σχέση με το 2001. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει ένα πρόγραμμα όταν υποβληθεί εμείς δίχως άλλο θα το προωθήσουμε. Διατυπώθηκε μία ερώτηση εθνικού χαρακτήρα θα έλεγα περισσότερο. Ο συνάδελφος ρώτησε τι έχουμε σκοπό να κάνουμε με την ε, ε, σε ό,τι αφορά ε, την διαφορά που παρατηρείται στις γραμμές ε, το τρένο στην Ιβηρική Χερσόνησο και σε άλλες χώρες. Θα ήθελα τη, η διαφορά αυτή και στην Ισπανία να είναι ίδια με αυτή που γίνεται αποδεκτή στους σιδηροδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως αυτό κοστίζει. Θα ασχίσουμε πιέσεις και δίχως άλλο είναι στόχος μας να το επιτύχουμε μη μου κάνετε άλλη ερώτηση για τους μεσογειακούς διαδρόμους. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που τόνισα ότι είναι ένας από τους στόχους μας. Δηλαδή μεταξύ των προτεραιοτήτων να συμπεριληφθεί και αυτό το θέμα των ε, μεσογειακών διαδρόμων. Πιστέψτε με, το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα θα πρέπει να ορίσουμε την μεθοδολογία η οποία θα διέπει τις μελλοντικέ μας εργασίες για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν αυτοί οι διάδρομοι. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσει να οριστεί η μεθοδολογία αυτή. Αν τα καταφέρουμε όλα τα υπόλοιπα θα είναι πολύ πιο εύκολα από αυτή την άποψη. Για μία ακόμα φορά θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ απόλυτα με την παρέμβαση που έκανε ο κ. Δεγκράντες. Ενημέρωση των ε, ταξιδιωτών. που ταξιδεύουν με το αεροπλάνο. Όπως γνωρίζετε, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν αναλάβει να αναπτύξουν δράσεις στα πλαίσια προγραμμάτων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Το πρόγραμμα υπαριθμών 3, υψηλή ταχύτητα, πρωταρχικός άξονας, ε, ε, Γάγια, Φιγκέρας, Περπινιών, ε, Ύστερα Σίνες, Αλχεσίρας, Μαδρίτη, Παρίσι που αποτελεί μέρος του, δια, του άξονα που περνάει από τα Πυρηναία Όρη. Πρόγραμμα υπαριθμών 19. Εκεί ε, συνεργαζόμαστε στενά με τη Γαλλία. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις με τη χώρα αυτή και υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία για να μπορέσουμε να κινηθούμε με όσο γίνεται πιο γοργούς ρυθμούς. Χαίρομαι, υπογραμμίζω, χαίρομαι για, για την απόφαση που υιοθετήθηκε για ένα νέο Ευρωπαίο συντονιστή που θα ασχολείται με το PP3. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω για το sd 3 Θα ήθελα για το, το 16 θα πρέπει επίσης να συντονιστεί από τον κύριο Σέκη έτσι ώστε να υπάρξει μία σαφέστερη άποψη για τους διαδρόμους στους οποίους ανέφερα. Το, το είπα ήδη στον ε, Επίτροπο Ταγιάννη και τώρα έχω σκοπό να πείσω τον Επίτροπο Κάλλας για να υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ των τριών διαδρόμων. Σε ό,τι αφορά τους, τα ηλεκτρονικά αρχεία των ε, φορτηγών σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουμε. Θα δημιουργηθεί αυτό το αρχείο τα επόμενα χρόνια. Θα πρόκειται για εθνικά αρχεία, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους. Η κρίση της εσωτερικής ναυσιπλοείας είναι ένα θέμα. Λαμβάνω υπόψη τα, τους προβληματισμούς που διατυπώσατε. Ε, θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το είχα σκεφτεί πριν από τη συνεδρίαση αυτή. Θα, θα ε, απαντήσω σε κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για τις απαντήσεις του στα ερωτήματα. Είχα πει στην αρχή ότι οι συνάδελφοι μερικές φορές ε, κάνουν δύσκολες ερωτήσεις και νομίζω ότι το κάνανε αυτό σήμερα. Επίσης πάντα θεωρούσα ότι ένα μειονέκτημα των Υπουργών Μεταφορών εδώ είναι ότι η Επιτροπή μας γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε καλά κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προτεραιότητες και τους στόχους σας. Και βεβαίως όπου μπορούμε Ευχαριστώ. θα συνεργαστούμε μαζί σας προκειμένου να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία που θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε τις μεταφορές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμευόμαστε λοιπόν απέναντί σας να συνεργαστούμε μαζί σας όπου είναι δυνατόν για την εκπλήρωση των στόχων της Προεδρίας σας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε που απαντήσατε και όλα τα ερωτήματά μας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους που με βοήθησαν προκειμένου να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, ειδικά τα δύο μέλη που απέσυραν τις ερωτήσεις σας. Και να υπενθυμίσω στα μέλη ότι στις 3 το απόγευμα θα υποδεχθούμε στην αίθουσα 5G3 Υπουργό Τουρισμού. 5G3. Θυμηθείτε να πάρετε κοντά σας